Uh, and Lamberts, would you like to possibly, please, very nicely, please? Um, take a seat. Sorry to break up your conversation. Yesterday after... Καθίστε παρακαλώ. Χθε αρχίσαμε 10 λεπτά αργότερα και ε, μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο σημείο είχαμε καθυστερήσει μισή ώρα, άρα ουσιαστικά δεν το καλύψαμε και έπρεπε να το συζητήσουμε και σήμερα. Γι' αυτό θα προσπαθώ πραγματικά να ξεκινάω από σήμερα πραγματικά στην ώρα μας. Να ξεκινάμε. Αυτή είναι η προειδοποίησή μου. Θα το προσπαθήσω, παρότι δεν το συνηθίζω. Σε ό,τι αφορά τα γεωσκοπικά δεδομένα, για εμπορικού λόγου, Γέννη Νίλσεν είναι ο εισηγητή μα η μελέτη αντικτύπου που θα μας παρουσιάσει η Επιτροπή από πιο συγκεκριμένα εκπρόσωπο θα γίνει παρουσίαση από τον κύριο Αγκόστο Γκονζάλες Ερνάντες. Καλώς ήρθατε, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Αγκόστο Γκονζάλες Ερνάντες, πολύ σωστά. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μα. Θα ήθελα να σα τονίσω λοιπόν αυτό το οποίο εμείς ε, θεωρούμε ότι είναι το σημαντικό μήνυμα αυτής της μελέτη αντικτύπου. Νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα γεωσκοπικά δεδομένα και υπηρεσίες ε, είναι σημαντικά για το περιβάλλον, τον χωροταξικό σχεδιασμό, τη γεωργία, τη διαχείριση φυσικών πόρων, τη διαχείριση καταστροφών, την άμυνα, την ασφάλεια. Μικρός είναι ο τομέας, ε, οι επιχειρήσεις δηλαδή οι οποίες δραστηριοποιούνται εν γέννη ε, σε αυτό το τομέα είναι γύρω στις 300 και κάνουν διάφορα πράγματα. Ο αριθμός τώρα των επιχειρήσεων που μας αφορούν πιο άμεσα είναι 100 περίπου τον αριθμό και είναι εταιρείε αυτές οι οποίες χρησιμοποιούν δεδομένα γεωσκοπικά για την παραγωγή ε, χαρτών, για χαρτογραφικές υπηρεσίες και τα σχετικά. Απασχολούν συνολικά οι 300 επιχειρήσει 5.000 περίπου άτομα, μεταξύ δε των εταιριών αυτών το 99% η συντριπτική τους ε, πλειοψηφία είναι μικροεπιχειρήσεις και το 67% πολύ μικρές επιχειρήσεις, πολύ μικρής κλίμακας, δηλαδή με 10 ή λιγότερους εργαζομένους. Αυτές είναι σημαντικές πληροφορίες, διότι μπορούμε να επηρεάσουμε αυτές τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και να δούμε τι μπορούμε να έχουμε από πλευράς πληροφοριών, ένας ε, πολλά υποσχόμενος τομέας. 700 εκατομμύρια έσοδα αυξάνονται και οι πωλήσει δεδομένων Τη τάξη του 7% ετησίως, καλό αυτό, αλλά όχι τόσο όσο με αυτά τα οποία συμβαίνουν στις ΗΠΑ όπου έχουμε ποσοστά ανάπτυξης τη τάξη του 9%. ή 19% δεν ήταν σαφές. Τώρα, τι γίνεται με τα δορυφαρικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης. Πώς γίνεται η διανομή τομεί τομείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Μπορεί να είναι λίγες επιχειρήσεις οι οποίες ε, κερδίζουν τα πιο πολλά χρήματα. Τέλος πάντων, ποιο είναι τώρα το θέμα, ποια είναι η ουσία. Τα δορυφικά δεδομένα υψηλή ανάλυσης ελέγχονται από τις κυβερνήσεις. Όποτε υπάρχει ένα δορυφορικό σύστημα που μπορεί να παράγει υψηλή ποιότητα τέτοια δεδομένα υψηλή ανάλυση, πρέπει οι εθνικέ αρχέ να τα ελέγχουν λόγω των προφανών ανησυχιών ασφάλεια. Δηλαδή, κανεί βλέπει πράγματα με πολύ μεγάλη ευκρίνεια. Υπάρχει λοιπόν η ανησυχία ότι κάποια από αυτά δεν θα έπρεπε να τα βλέπει κανεί. Και αυτό ισχύει τόσο εντό όσο και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, ούτω εχόντων των πραγμάτων και για του σκοπού τη μελέτη αντικτύπου, Κάναμε μια ανάλυση των χαρακτηριστικών των συστημάτων αυτών που έχουμε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρία κράτη-μέλη, ίσως και ένα τέταρτο, με δορυφικά σύστηματα υψηλής ανάλυσης και μέτρα ελέγχου για τα δεδομένα που μπορούν να συλλέγουν τα συστήματα αυτά. Κατά βάση δεν υπάρχει μια κοινή συμφωνία για το τι εστί υψηλή ανάλυση, η υψηλή ευκρίνεια. Οι επιχειρήσεις σήμερα έχουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ότι δεν γνωρίζουν ουσιαστικά τι είναι αυτά τα δεδομένα υψηλή ανάλυση, άρα δεν είναι και βέβαιε επιχειρήσει ε, όταν θέλουν να αγοράσουν τέτοιου είδου δεδομένα. Ότι ε, θα υποβληθούν ή δεν θα υποβληθούν σε ελέγχου. Δεν είναι βέβαιο αυτό δεν το γνωρίζουν. Επίση, ξέρουμε ότι τα εφιστάμενα συστήματα χαρακτηρίζονται και από διαφορετικά επίπεδα διαφάνεια. Έλεγχοι ναι, μεν υπάρχουν, όμω οι επιχειρήσει στον τομέα αυτό δεν γνωρίζουν κατά ανάγκη πότε θα γίνει ο έλεγχο και με ποια κριτήρια. Δηλαδή, αν κάποιο θέλει να αγοράσει υψηλά, υψηλής ανάλυση δορυφορικά δεδομένα, δεν ξέρει αν αυτά θα είναι ευαίσθητα από θέματα ασφάλειας ή όχι, γιατί τα κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται δεν είναι δημοσιοποιημένα, δεν είναι γνωστά. Η πρόσβαση τώρα στα δεδομένα. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει έλεγχο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι μπορεί να υπάρξει σε ένα άλλο κράτο μέλο ο έλεγχο. Α πούμε ότι είστε μια μικρή επιχείρηση, αγοράζετε από πάροχο δεδομένων σε ένα συγκεκριμένο κράτο μέλο τα δεδομένα αυτά. Γίνονται οι έλεγχοι, αλλά δεν αποτρέπει σήμερα ε, κάτι, ε, ένα άλλο κράτος μέλος να προβεί σε κάποιους έλεγχους. Δεν υπάρχει κοινή προσέγγιση στα θέματα αυτά. Άρα δεν υπάρχει και ελεύθερη κυκλοφορία δορυφορικών δεδομένων υψηλή ανάλυση Το ίδιο ισχύει. και στα δεδομένα μικρής ή μεσαίας ευκρίνειας. Υπάρχουν δηλαδή αυτά τα δεδομένα που δεν θεωρούνται ευαίσθητα πολύ ασφάλεια, αλλά ότι και και αυτά υπάρχει εγγύηση ότι μπορεί να είναι η διανομή τους ελεύθερη και η κυκλοφορία τους ελεύθερη. Όταν αναλύαμε την κατάσταση, προέκυψε και το εξή. Επειδή τα εθνικά συστήματα που υπάρχουν σήμερα έχουν σχεδιαστεί για εθνικού σκοπού, φαίνεται να επηρεάζεται ε, ο εντοπισμός των εταιριών. Όπως μας είπε ο εξωτερικός σύμβουλος, το 60% των εταιριών είναι σε τρία κράτη-μέλη ουσιαστικά. Και υπάρχει και το σύστημα ελέγχου για την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα υψηλής ανάλυσης. Ποια είναι η ουσία τώρα. Ποια είναι τα δεδομένα, ποιο είναι το ποσοστό των δεδομένων που ελέγχονται. 1% των δεδομένων ψηλής ανάλυσης είναι περιορισμένα ή ελέγχονται, έτσι μας είπε ο εξωτερικός σύμβουλος. Πολύ μικρό το ποσοστό. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι υπάρχουν διαφορές μεταχείρισης των δεδομένων ανάλογα με το κράτος μέλου. Αυτό δεν δημιουργεί ουσιαστικά πρόβλημα, αφού είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό αυτών των δεδομένων. 1% όπως είπα. Δεν έχει και τόση μεγάλη σημασία λοιπόν. Θέλησαμε να δούμε όμως αν ισχύει αυτό ή όχι γι' αυτό. Και διεξαγάγαμε μια διαβούλευση, ήρθαμε σε επαφή με τη βιομηχανία, αλλά κάναμε και μια ηλεκτρονική έρευνα για τις επιχείρησεις που θεωρούμε ότι ε, έχουν να κάνουν στην επιχειρηματική του δραστηριότητα με δεδομένα υψηλής ανάλυσης και συγκεκριμένα 47 εταιρείες από την ΕΡΣΚ. Απάτησαν 20. Μπορεί να σας φαίνεται μικρός αριθμός. Αλλά αν σκεφτείτε ότι συνολικά όλες οι εταιρείες οι οποίες εργάζονται στο τομέα αυτό είναι 120, νομίζω ότι είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό το δείγμα. Και σε αντίθεση με αυτό που θα μπορούσε να αναμένει κανείς περισσότερες αντιμετώπισαν προβλήματα στην πρόσβαση δεδομένων οι 15 στις 20 8 είπαν έχουμε δυσκολίες αλλά δεν γνωρίζουμε από πού προέρχονται θα μπορεί να οφείλονταν στον καιρό δεν ξέρω εγώ που αλλού τέσσερις εντόπισαν δυσκολίες ή τέλο πάντων να μας έδωσαν άλλου λόγους. Ναι, μεν είναι μικρά τα απόλυτα νούμερα, όμως υπάρχει ένα σαφές ποσοστό εταιριών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την πρόσβαση τέτοιων ε, δεδομένων, για τον τομέα της τηλεανείχνευσης συγκεκριμένο από την ΕΡΣΚ. Είπαμε ότι δεν ε, είναι σαφές τι σημαίνει υψηλή ανάλυση. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Και το θέμα το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει ένα διαφανέ σύστημα για να γνωρίζουν επιχειρήσεις με τι κριτήρια αποφασίζεται ε, αν ένα δεδομένο θεωρείται ευαίσθητο από πλευρά ασφάλεια ή όχι. Ρωτήσαμε, κάναμε κάποιες ερωτήσεις για το θέμα αυτό και εδώ η συντριπτική πλειοψηφία ήταν υπέρ του να υπάρχει αυτό το διαφανέ σύστημα 12 στις 20 εταιρείε μα ε, αποφάσισαν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια, ένας κοινό ορισμός, μια κοινή συνεννόηση για το TST δεδομένου υψηλή ανάλυσης και 14 στις 20 είπαν ότι θα ήταν καλό να υπάρχουν κοινά κριτήρια ώστε να μπορούν να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις πότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ελεγχθούν ή όχι τα δεδομένα. Από το πρίσμα όλων αυτών των στοιχείων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στη μελέτη αντικτύπου να αναπτυχθεί μια προσέγγιση η οποία θα θεσπίζει κατόφλια που θα ορίζουν τα δορυφικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης, οπότε θα υπάρχει ε, μια κοινή κατανόηση όχι μόνο του τι είναι, αλλά και του τι δεν είναι δορυφικό δεδομένο ψηλής ανάλυσης. Και επομένως, επομένως λέγω, θα δίνεται ένας ορισμός με τον τρόπο αυτό, ώστε θα αποκλείονται από ελέγχους ασφάλειας τα δεδομένα μικρής μέσης ευκρίνειας. Άρα, με το σύστημα αυτό θα ξέρουμε τι ενδεχόμενα μπορεί να ελεγχθεί, αλλά και τι δεν θα ελέγχεται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις. Δεύτερο στοιχείο της μετροπαθούς αυτής προσέγγισης. Θα θεσπιστούν Παρόμοιε όχι ταυτόσιμε, αλλά παρόμοιε διαδικασίε ελέγχου. Έτσι επιχειρήσει θα μπορούν να γνωρίζουν τα αιτήματα για δορυφορικά δεδομένα υψηλή ευκρίνεια. Πώς θα ε, αντιμετωπίζονται και πόσο χρόνο θα χρειάζεται μέχρι ότου έχουν ένα αποτέλεσμα. Αν πρέπει να υπάρξει έλεγχο αυτών των δεδομένων. Τέλος. Η προσέγγιση που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να εξασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που δεν είναι υψηλή ανάλυση μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Αυτά που είναι υψηλή ανάλυση όμω δεν θα υποβάλλονται σε διπλού ελέγχου. Και αν δεν ελέγχονται ή αν έχουν ελεγχθεί άπαξ, θα μπορούν πλέον να κυκλοφορούν ελεύθερα. Δύο λόγια τώρα για τον αντίκτυπο. Αναλύσαμε τα προβλήματα, προτείναμε έναν τρόπο αντιμετώπιση των προβλημάτων, αναλύσαμε τους αντικτύπους, τις επιπτώσεις. Αξιολόγηση τώρα και ποσοτικοποίηση του οικονομικού αντικτύπου. Πολύ δύσκολο εγχείρημα. Και όπως είπα, στην αρχή αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μιλάμε για πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις. Εκτός του ερωτηματολογίου ήρθαμε και σε άμεση επαφή με τις επιχειρήσεις αυτές, ζητώντας τους αν είναι δυνατόν να μας ποσοτικοποιήσουν τον αντίκτυπο μιας αλλαγή στην κατάσταση και κατά βάση μας είπαν ότι δεν έχουν τα μέσα ή τους πόρου προ κάτι τέτοιο. Άρα με δικές μας προσπάθειες και του Εξωτερικού Συμβούλου ε, δεν μπορέσαμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Είναι εύκολο βέβαια από την ανάλυση που έγινε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι αν δεν κάνουμε τίποτα τα προβλήματα που εντοπίσαμε θα επιμείνουν. Επίσης, ε, ο σύμβουλος υποστηρίζει ότι αν αφήσουμε την κατάσταση αμετάβλητη, οι μεγάλες πιθανότητες είναι. Ναι, μεν θα αναπτυχθούν και άλλα δορυφορικά συστήματα υψηλή ανάλυση, άρα και περισσότερα κράτη-μέλη θα ε, δικά του συστήματα, θα, έχουν, θα έχουμε απόκληση ε, στι διάφορε προσεγγίσεις, άρα ε, και μεγαλύτερη απόκληση ακόμα. Άρα υπάρχει κίνδυνο να χάσουν οι πελάτες οι επιχειρήσεις. Δεν θα μπορούν να παραδίδουν εγκαίρως τα προϊόντα του προϊόντα τους και να πούν στον πελάτη ότι μπορώ να προγραμματίσω εκ των προτέρων και να σου εγγυηθώ ότι θα έχεις αυτά τα δεδομένα όταν τα χρειάζεσαι. Καταλήξαμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι επειδή δεν υπάρχει κοινό ορισμός ή κοινή προσέγγιση για κάποιες διαδικασίες και επειδή δεν έχουμε και κάποιο νομοθέτημα, δεν έχουμε πολλά δηλαδή πράγματα στη διάθεσή μας, αλλά μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια θετικά συμπεράσματα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίε έχουν δεσπόζουσα θέση ε, σε αυτό το τομέα τη παρατήρηση τη γη, έχουν νομοθεσία για τα δεδομένα υψηλή ανάσα το 1988. Εμείς έχουμε μείνει δεκαετίες πίσω. Ε, και υπάρχει το θέμα της ισότιμης πρόσβασης ε, στα δεδομένα υψηλής ανάλυσης. Βέβαια, στην ΕΠΑ υπάρχει και επιθετική πολιτική από πλευρά κυβέρνηση και αυτό ωφελεί τι επιχειρήσει. Οι επιχειρήσει όμω δεν έχουν να αντιμετωπίσουν εκεί διαφοροποιημένα συστήματα, αποκλίνοντα συστήματα. Η κατάσταση εδώ είναι πολύ διαφορετική. Αυτά έχω να πω προς το παρόν. Ευχαριστώ. Thank you. Jens. Ευχαριστούμε πολύ. Γιάννης Νίλσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις παρατηρήσεις της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζουμε ότι προσπαθεί να επιτύχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα με αυτή την προσπάθεια και γι' αυτό είναι και μια πολύ σημαντική ρυθμιστική πρόταση. Ενδιαφέρον είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να ρυθμίσει τον συγκεκριμένο τομέα. Αυτό που πρέπει να αποφύγουμε εμείς είναι να συνυπάρχουν ταυτόχρονα διαφορετικοί εθνικοί κανόνες, διότι αυτό θα δυσχεράνει την εφαρμογή του κανονισμού. Πρέπει να λύσουμε συγκεκριμένα προβλήματα και όπως υπόθηκε υπάρχουν τρία μόνο κράτη-μέλη τα οποία έχουν προβεί σε αυτές τις ρυθμιστικές ενέργειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίλησε για έναν κατάλογο τη δημιουργία ενός καταλόγου και εμείς θα θέλαμε να μάθουμε πώς ακριβώς σκοπεύει να επιλύσει αυτά τα προβλήματα. Είναι γνωστή η κατάσταση που ε, επικρατεί στο Συμβούλιο, είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί, περιμένουν περαιτέρω αναλύσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όταν φτάσουν αυτές οι αναλύσεις πρέπει και εμείς να είμαστε σε ετοιμότητα. Εγώ Κρατώ ανοιχτό μυαλό, είμαι έτοιμος να ακούσω όλες τις ε, συνεισφορές, να διαβάσω την εκτίμηση αντικτύπου και φυσικά ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για το τι θα γίνει και σε αυτήν εδώ την Επιτροπή και στα άλλα θεσμικά όργανα. Όσον αφορά, με τις, διαβουλεύσεις με τις ε, ε, εταιρείε, από ό,τι καταλαβαίνω δεν έγιναν άμεσες διαβουλεύσεις και θα έπρεπε πιστεύω να γίνουν, διότι υπάρχουν πολλέ εταιρείε οι οποίες έχουν δείξει ενδιαφέρον και έχουν μάλιστα εμπειρία η οποία θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη. Οι εταιρείε αυτές ασχολούνται με την πρακτική εφαρμογή αυτών των γεωσκοπικών δεδομένων Και εδώ συζητούμε για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως χρειάζεται προσοχή, διότι 12 εταιρείες στην Ευρώπη, η συντριπτική πλειοψηφία από αυτές απάντησε, 7 απάντησαν από τους 12 που ερωτήθηκαν και τα πράγματα είναι κάπως δύσκολα, διότι η συντριπτική πλειοψηφία μπορεί να ακούγεται ωραία σαν έκφραση, όμως πρέπει να δείξουμε προσοχή. Όμως, όπως είπα, περιμένω να συνεχιστεί η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βανίστελ Ρόι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που άκουσα για τις εξελίξεις στον κλάδο. Πιστεύω πως η Επιτροπή μας πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι εάν πρέπει να κάνει κάτι, πρέπει να το κάνει τώρα, διότι έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε στις εταιρείε τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες γι' αυτό και δεν πρέπει να τις χάσουμε. Οι Αμερικάνοι, για παράδειγμα, πριν δέκα χρόνια δεν είχαν μεγάλη αγορά και τώρα υπάρχει κατακαιρματισμός αυτής της αγοράς. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν καινούργιες ευκαιρίες για τις μικρές εταιρείες ειδικότερα, έτσι ώστε αυτές να αναπτυχθούν και να μεγαλώσουν. Μας είπατε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες, όμως εγώ πιστεύω πως χρειαζόμαστε και δράση. Τα πρότυπα για την κινητή τηλεφωνία, για παράδειγμα, στην Ευρώπη ήταν κάτι που μας έδωσε τον ηγετικό ρόλο παγκοσμίω. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει εμείς εδώ σε αυτήν την Επιτροπή να ασχοληθούμε με πράξεις. Και κοιτάζω εσάς κυρία Πρόεδρε, διότι ξέρω πως έχουμε ένα θέμα αρμοδιότητας το οποίο πρέπει να διαπραγματευτούμε. Θα πρότεινα λοιπόν να κοιτάξουμε και άλλες περιπτώσεις όπου έγιναν λάθη. Να δούμε ακριβώς τι συνέβη και να το χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να θέσουμε τη νέα μας πορεία. Διότι εντάξει, οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικός παίκτη, όμως πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τη μελέτη και ας πάρουμε τον ηγετικό ρόλο εδώ στην Επιτροπή ΙΝΚΟ και ας δούμε τις ευκαιρίες που μπορούν να μας ανοιχτούν, διότι πραγματικά υπάρχει μεγάλο δυναμικό. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για αυτή τη μελέτη και πραγματικά πιστεύω πως έχει έρθει η ώρα να πιάσουμε δουλειά και να μην αναβάλουμε τα πράγματα για το μέλλον. I'm uh, content to just... Όχι, όχι, προτιμώ να ακούσω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συνάδελφοι, κυρία Γκέπχαρτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον και σημαντικό το θέμα αυτό. Διότι αφορά άμεσα την εσωτερική αγορά και είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Πιστεύω πως ε, ο Γένς είχε δίκιο με το ότι πρέπει να πάμε μπροστά. Πιστεύω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ίδιο είπε. Χρειάζεται όμως προσοχή. Πρέπει να βρούμε τις σωστές ε, λύσεις, τον σωστό τρόπο για να προχωρήσουμε. Ε, έχω κάποιες ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι θα ήθελα να μάθω λίγα περισσότερα για το γιατί η πρόταση έχει τη μορφή που έχει. Λέτε λοιπόν στην αρχή των αιτιολογικών σκέψεων ότι υπάρχει ανάγκη για ευρωπαϊκή ρύθμιση. Όμως όταν βλέπω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπω ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ρύθμιση, υπάρχουν 28 διαφορετικές ρυθμίσεις των κρατών μελών. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω ε, είναι το αν πραγματικά είναι εφικτή μια ευρωπαϊκή, πανευρωπαϊκή ρύθμιση. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και θα μπορού, και όπως λέει και ο αρμόδιος επίτροπος κύριος Ότινγκερ, χρειάζονται ευρωπαϊκές λύσεις και δεν γίνεται λοιπόν να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις ε, εθνικές ρυθμίσεις διότι η εσωτερική αγορά δεν έχει σύνορα και είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το δεύτερο που θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με δορυφορικά δεδομένα και η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ ώστε τα δεδομένα που λαμβάνουμε προέρχονται από πάρα πολλούς ε, άλλους ε, τομείς και πιστεύω πως η τεχνολογία μας προσπερνά. Υπάρχουν δεδομένα δηλαδή που δεν παίρνουμε μόνο από δορυφόρους αλλά και από μη επανδρομένα οχήματα, σκάφη και πρέπει πραγματικά να ασχοληθούμε με την προστασία της ε, ιδιωτικής σφαίρας των πολιτών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικότερο από τα δορυφορικά δεδομένα καθ' αυτά. Ας μην τρέχουμε συνέχεια πίσω από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Έχετε λοιπόν ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιες προτάσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Στην εσωτερική αγορά πραγματικά πρέπει να κοιτάζουμε την τεχνολογία του αύριο και να σκεφτόμαστε με γνώμονα αυτήν και όχι με την τεχνολογία του χθες. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να κάνει ερωτήσεις. Θα ήθελα και εγώ να συνεχίσω την ερώτηση του κύριου Λάμπερτς και να πω ότι ενδεχομένως να υπάρξει πρόβλημα αρμοδιότητας με την Επιτροπή Ήτρε. Αλλά το θέμα αυτό θα επιληθεί στη διάσκεψη των Προέδρων. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία έχουν ανατεθεί σε εμά και κάποια που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή ΙΤΡΕ. Θα ξεκαθαριστεί όμως. Όπως και να έχει, αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι καταρχάς ότι το θέμα αυτό είναι περίπλοκο και υπάρχει για το θέμα του κόστους και αυτό είναι κατανοητό, διότι υπάρχει μεγάλο κόστος το να στείλει ένα δορυφόρο στο διάστημα. Μόνο τρει χώρε το έχουν καταφέρει και υπάρχουν κάποιες άλλες χώρε που το κοιτάζουν. Ο δορυφορικός, ε, ο τομέας της δορυφορικής τεχνολογίας είναι ένας τομέας ο οποίος μεγαλώνει, μεγαλώνει ταχύτατα και υπάρχει επιθυμία να αυξηθεί η ευρωπαϊκή παρουσία. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ερωτήσω τι άποψη έχουν οι εκπρόσωποι του κλάδου της δορυφορικής βιομηχανίας, εάν γνωρίζετε φυσικά. Εάν σκεπτικό μας είναι τα δορυφορικά δεδομένα να εναρμονιστούν στην ευρωπαϊκή προσέγγιση, και γνωρίζω φυσικά ότι υπάρχουν μεγάλες ευαισθησίες σχετικά με τα δεδομένα και σε πολλούς τομείς, και ακριβώς επειδή οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν τη δική τους πολιτική όσον αφορά τη χρήση δεδομένων για λόγους ασφαλείας και ε, για άλλους σκοπούς, ε, δεν εξυπακούεται ότι και εμείς θα ακολουθήσουμε την ίδια πολιτική με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ξέρω λοιπόν ότι είναι ευαίσθητο το θέμα και μπορώ να καταλάβω γιατί Κάποια κράτη-μέλη έχουν ανησυχίες για τα θέματα ασφαλείας. Αυτό το είδαμε και στη συζήτηση για τα συστήματα και τα δίκτυα ασφαλείας. Όλα φαίνονται πιο εύκολα βέβαια στο χαρτί, όμως πραγματικά είναι πολύ ευαίσθητα θέματα αυτά. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι τι άποψη έχουν οι ίδιοι εκπρόσωποι του κλάδου της ορφορικής βιομηχανίας και έπειτα γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα Γαλιλαίος και Κοπέρνικος. Προσπαθούμε να έχουμε τους ίδιους κανόνες εκεί, διαφορετικούς. διότι εγώ βρίσκομαι πολλές ομοιότητες ε, στα θέματα που αφορούν τα δεδομένα. The Θα μπορούσε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σωστά τα είπατε. Πέραν των τριών κρατών μελών που ήδη έχουν δυνατότητε ε, και προβλέπεται από τη δικαιοδοσία τους, ε, έχουμε άλλες δύο χώρες που ετοιμάζονται σε ό,τι αφορά τη διαβούλευση Ίσως να ήταν λίγο υπερβολή όταν είπα για τη συντριπτική πλειοψηφία σε σχέση βέβαια αν το συγκρίνει κανεί με, ε, με τον αριθμό το συνολικό. Απλά λέω για αυτούς που απάντησαν, η πλειοψηφία αυτών που απάντησαν. Τώρα όμως ε, που έχει δημοσιοποιηθεί οδηγία, διεξάγουμε και μια ακόμη έρευνα, την οποία την δρομολογήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και θα έχει ολοκληρωθεί την Κυριακή που μας έρχεται. Και πάλι βέβαια δεν είχαμε μαζική ανταπόκριση, 22 απαντήσεις λάβαμε. Το ενδιαφέρον στοιχείο, προκαταρκτικά, που μπορώ να σας πω, είναι ότι είναι ακριβώς προς την ίδια κατεύθυνση απαντήσεις και το ενδιαφέρον είναι ότι είναι άλλες εταιρείε. Είχαμε δηλαδή μια πρώτη έρευνα για την προετοιμασία της μελέτης αντικτύπου. Τώρα έχουμε μια άλλη έρευνα για να ακούσουμε τι θέλει να μας πει ο κλάδος και περιλαμβάνονται εδώ οι ε, πάροχοι υπηρεσιών δορυφορικών. Θα δούμε τι έχουν να μας πούν και αυτοί και επομένως πρόκειται αυτή τη φορά για διαφορετικές εταιρείε. Οι απαντήσεις που δίνουν όμως είναι προς την κατεύθυνση και αυτό είναι χρήσιμο σε σχέση με αυτό που επιθυμούμε να κάνουμε. Περιορισμένο είναι σίγουρα το πεδίο Συμφωνώ, ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερες. Πιστεύω όμω ότι πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα. Κατέληξε η Κομισιόν στο συμπέρασμα ότι καλό θα ήταν να εντοπίσουμε πού υπάρχει το πρόβλημα με την πρόσβαση των δεδομένων. Και γι' αυτό έχουμε αυτή την συγκεκριμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση που ταυτόχρονα όμως σέβεται και τι αρμοδιότητε των κρατών μελών, που είναι αποκλειστικές ε, οι αρμοδιότητες για το τομέα τη ασφάλεια. Ναι, μεν λοιπόν έχουμε τον κοινό ορισμό ε, της ψηλής ανάλυσης και έχουμε κάποιε παρόμοιε διαδικασίες για την οδέσμευση δεδομένων λόγω ασφαλεία. Δεν επιβάλλουμε τίποτα στα κράτη-μέλη, δηλαδή δεν επιβάλλουμε συγκεκριμένα κριτήρια, προτείνουμε όμως ε, να εγκριθεί μια παρόμοια προσέγγιση η οποία θα διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων. Δεν θα έλεγα βέβαια ότι θα έχουμε 20 κανόνες, κάτι καλύτερο θα πετύχουμε. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να αποκτώνται αυτά τα δεδομένα υψηλής ανάλυσης όπως είναι τα τηλεκατευθυνόμενα, τα drones. Ξέρετε όμως υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ δορυφορικών δεδομένων και τηλεκατευθυνόμενων. Εγώ διαφωνώ ότι είναι τεχνολογία του παρελθόντος ε, ε, οι δορυφόροι του μέλλοντος θα τη χαρακτηρίζω εγώ. Αλλά τέλος πάντων ε, το, αντιμετωπίζουμε το ζήτημα αυτό, την απόκτηση των δεδομένων από το διάστημα, με ε, τηλεκατευθυνόμενα που αν δεν θέλουμε να πετούν πάνω από κάποια συγκεκριμένη περιοχή ε, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τρέψουμε την πτήση αυτό το τηλεκατευθυνόμενο, ενώ οι δορυφόροι δεν έχουν τέτοιο περιορισμό, διότι είναι σε τροχιά γύρω από τη γη συνεχώς και πηγαίνουν παντού κατά κάποιο τρόπο. Μπορούν επομένω να πάρουν στοιχεία. Τα αεροπλάνα ή τα τηλεκατευθυνόμενα ε, μπορεί να μην μπορούν να πετάξουν παντού. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε και με το θέμα αυτό βέβαια. Όμως, για το διαστημικό τομέα λέω, υπάρχει μεγάλη ανάγκη να παρέμβουμε στο τομέα αυτό. Τέλο, κύριε Πρόεδρε, ρωτήσατε γιατί αποκλείουμε ή εξαιρούμε αν θέλετε καλύτερα το Κοπέρνικος. Η οδηγία αυτή απευθύνεται στα κράτη-μέλη. Ο Κοπέρνικος υπάρχει, διέπεται από κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Με αυτόν τον κανονισμό ορίζονται όλα, όλες οι πτυχές. Υπάρχει μια κατεξουσιοδότηση πράξη της Κομισιόν για δεδομένα τα οποία είναι πολύ παρόμοια να μην πω ταυτόσιμα σχεδόν, με την προσέγγιση της οδηγίας. Η προσέγγιση με το κοπέ, για το ό,τι αφορά δυνητικά ε, δορυφορικά δεδομένα υψηλή ευκρίνεια η ανάλυση, αυτό ρυθμίζεται από την κατεξοδότηση πράξη της Κομισιόν. Για τα ειδικά δεδομένα του Κοπέρνικου. Παρόμοια, επαναλαμβάνω πολύ παρόμοια είναι η προσέγγιση όμως με αυτή που υιοθετούμε στην οδηγία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ θα μου άρεσε να γνωρίζω ποιες είναι οι διαφορές. Ποια είναι η διαφορετική προσέγγιση ε, για τα στοιχεία που συλλέγονται από τα κράτη-μέλη έναντι των στοιχείων που συλλέγει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γέννη, θα ήθελα να ξαναπάρει το λόγο, γιατί φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την αγγλική μετάφραση. Αγγλική μετάφραση έχουμε. Oh, I'm getting, I'm εγώ ακούω δανέζικα. Πάντως. Ναι, ναι, κι εγώ. <coughs> Jens. Ωραία. Εγώ καταλαβαίνω λίγο τα δανέζικα, οπότε κατάφερα να παρακολουθήσω τη συζήτηση. Πάντως ε, να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση. διάφοροι συνάδελφοι επανέλαβαν τα όσα έλεγα και εγώ. Είναι αλήθεια πως ε, η αγορά δεν είναι όρημη και ότι υπάρχει η δυνατότητα να ε, φτιαχτεί μια ομοιόμορφη οδηγία μια ρύθμιση ομοιόμορφη για ολόκληρη την Ευρώπη. Βέβαια αυτή είναι η πρόκληση. Υπάρχουν ακόμα δυσκολίες που θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε, αλλά ε, πιστεύω πως και αυτές θα μπορούσα να τις συζητήσω με τους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να δούμε ποιες ε, εκθέσεις θα μας δοθούν καταρχήν από τη διάσκεψη των Προέδρων. Ωραία λοιπόν, θα ψηφίσουμε στις 9.45. Ε, um, and just so, uh, thank you members Σας ευχαριστώ που ήρθατε όλοι υπέροχα. Απλά να σας πω κάτι για να το ξέρετε. Χτες το απόγευμα αρχίσαμε 10 λεπτά αργότερα και μέχρι ότου να φτάσουμε στα διάφορα στην ατζέντα είχαμε καθυστερήσει μισή ώρα. Γι' αυτό έκανα την υπόσχεση σε όλους όσους ήταν σήμερα εδώ ε, από την αρχή. Θα προσπαθήσουμε από εδώ και στο εξή να ε, ακολουθούμε αυστηρά το χρόνο της σημερινή διάταξη. Έχουμε άλλο ένα λεπτό μέχρι ότου να ψηφίσουμε. Okay. So members who have um, not yet arrived have just been some time because Ωραία λοιπόν. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή να μιλήσει και νομίζω από ό,τι κατάλαβα η Ιταλική Προεδρία θέλει να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να πω και πολλά. Ε, βασικά να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στη σύνταξη της έκθεσης. Δεν ήταν εύκολη η έκθεση. Ξεκινήσαμε πριν από τρία χρόνια Όπως ξέρετε, είχαμε μια πρωτοβουλία ε, ε, μαζί με την Επιτροπή ε, Τραν. Ήταν πολύ εντατική η συνεργασία μας για τρία χρόνια και τώρα φτάνουμε στο τέλος αυτής της δουλειάς. Και θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλους τους συναδέλφους για την αποτελεσματική και παραγωγική συνεργασία. Να ευχαριστήσω και την Ιταλική Προεδρία που έθεσε ως προτεραιότητά της την έκθεση αυτή. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία και από τις δύο πλευρές. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι και πιστεύω πως η σημερινή ψηφοφορία σημαίνει ένα μέγα άλμα προς ασφαλέστερους δρόμους μπορούμε να αποδείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να, είναι, να λειτουργεί προς όφελος του Εβραίου κοινού. Σας ευχαριστώ και πάλι λοιπόν για τη στήριξή σας και νομίζω πως όλοι θα στηρίξουμε αυτή την έκθεση όχι μόνο σήμερα αλλά και σε ένα-δυο μήνες στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ. Ακούς, Βανέσα παλίλο από την Ιταλική Προεδρία. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους σας. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Σιρανόβα, τους ε, σκιώδεις εισηγητές για την εξαιρετική συνεργασία που διέκρινε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις που τελικά ολοκληρώθηκαν με την επίτευξη της συμφωνίας. Να ευχαριστήσω επίσης τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, τη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής ΙΜΚΟ, καθώς και όλους τους ε, υπαλλήλους του Κοινοβουλίου που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση, στην επίτευξη μάλλον αυτής της συμφωνίας. Και τέλος, ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διευκόλυνε τις διαπραγματεύσεις και την επίτευξη συμφωνιών για πολύ σημαντικά και δύσκολα θέματα. Είναι μια, ένα πολύ σημαντικό θέμα για τους Ευρωπαίους πολίτες που ασκεί και παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση των θανάτων και των τραυματισμών στα αυτοκινηστικά δυστυχήματα. Πρόκειται ένα σύστημα επίγουσας κλήσης με βάση το νούμερο 112 και θα είναι πιο εύκολο να καταγράψουμε συγκεκριμένους κώδικες, να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες βοήθειας, άμεσης της βοήθειας και να μειωθούν ε, τα μηνύματα SOS στους δρόμους. Ε, η επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωκοινοβούλιο σε αυτό το συγκοινωνισμό απετέλεσε ε, προτεραιότητα για την Ιταλική Προεδρία από την αρχή του εξαμήνου και σε αυτή την οπτική στο Συμβουλίο επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την έγκριση του και μάλιστα με τα χαρά μπορώ να σας ανακοινώσω ότι είμαστε σε θέση να υιοθετήσουμε πολιτική συμφωνία για αυτόν τον κανονισμό στις 17 Δεκεμβρίου κιόλας, ώστε ε, να έχουμε κοινή θέση για τον ε, Φεβρουάριο και να δώσουμε τη δυνατότητα να το εκφράσει την ψήφο του από το Μάρτιο του 2015 στην Ολομέλεια και να φτάσουμε στην δημοσίευση του σημαντικού αυτού ε, κανονισμού. Ευχαριστώ και πάλι όλους για τη συνεργασία και για την καρποφόρα συμφωνία που επιτεύχθη που είναι τόσο σημαντική. Σας ευχαριστώ. Um, Μιλάμε για μία ε, μονοψήφο τώρα θα ψηφοφορία για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, εκτός αν θέλει και κάποιος άλλος το λόγο. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, έχουμε έναν σοσιαλιστή παραπάνω. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. 30 in favor. 32 ψήφοι υπέρ, μία κατά, δύο αποχές. Σας ευχαριστώ πολύ. Okay. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και την διαπραγματευτική ομάδα. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, ο οποίος συνεργάστηκε και με δύο άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Um, Το επόμενο σημείο λοιπόν της ημερήσιας διάταξης ε, είναι μια παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με τις μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Είναι μια έκθεση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων η εισηγητής της Επιτροπής Νομικών Οποθέσεων Πασκάλ Τεγκράντες. Επίσης θα γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Απασχόλησης και η εισηγήτρια της δικής μας Επιτροπής είναι η Μαρλένε Μίτσι. Ο κύριος Κούρτς θα μας κάνει την παρουσίαση και τον καλωσορίζω στην Επιτροπή μας. Έχουμε και τις διαφάνειες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. Θα δώσω το λόγο λοιπόν αμέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Um, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και καλημέρα. Θα ξεκινήσω με το πλαίσιο της πρωτοβουλίας. Το 98% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αντιστοιχούν στο 65% των θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρουσία τους ε, τώρα και οι δυνατότητες που έχουν ε, δεν ε, έχουν ακόμη εξαντληθεί, άρα μπορούμε, έχουμε ακόμη μεγάλο δυναμικό. 2% των ΜΜΕ βλέπετε ότι επενδύουν στο εξωτερικό για τη δημιουργία παρατημάτων εκτός της έδρας της χώρας που έχουν την έδρα τους. Είναι χαμηλό το ποσοστό, πολύ χαμηλό και μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Πώς όμως. Λαμβάνοντας ιδίω υπόψη το γεγονός ότι το επιχειρηματικό πνεύμα στην Ευρώπη υπολείπεται κάπως αυτού άλλων ανταγωνιστών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλαμε λοιπόν, και αυτή είναι η ιδέα μας, να προσπαθήσουμε να απλουστεύσουμε τη ζωή των ΜΜΕ, να αναπτύξουμε περαιτέρω το επιχειρηματικό πνεύμα και να προσαρμοστούμε στην ψηφιακή εποχή. Αν ρωτήσετε νέους επιχειρηματίες τι θέλουν τελικά από το εταιρικό δίκαιο στην αγορά, γιατί υπάρχουν και άλλα προβλήματα βέβαια που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά μιλάμε τώρα για την πλευρά του εταιρικού δικαίου. Να έχουμε απαιτήσει και να έχουμε χαμηλό το ε, κεφάλαιο το αρχικό για να είναι ευκολή η δημιουργία επιχειρήσεων. Και υπήρξε και ένα μανιφέστο που έγραψαν οι επιχειρηματίες. Και μάλιστα αυτή που έχουν εταιρείε που δημιουργούν πάνω το 50% των θέσεων απασχόληση. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε χαμηλέ επενδύσει. Ε, μάλλον θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τι χαμηλέ επενδύσει, το ε, όχι τόσο λαμπρό επιχειρηματικό πνεύμα που βλέπουμε στην Ευρώπη. Είδαμε λοιπόν κάποιε δυνατότητε αυτή τη μελέτη αντικτύπου. Μία από αυτέ ήταν να δημιουργηθεί μια νέα νομική μορφή. Ένας νέος τύπος εταιριών ή ίσως να τροποποιηθούν οι φυστάμενοι τύποι εταιριών. Και αυτό θεώρησαμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχει ιστορία πίσω από το εταιρικό δίκαιο, έχουμε ε, το δίκαιο το εθνικό, έχουμε υπερεθνικά μορφές επίσης εταιριών, άρα είναι πολύ δύσκολο να διαπραγματευτούμε. Το Κοινοβούλιο πρέπει να σας πω ότι δεν συμμετέχει άμεσα σε τέτοιες διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου 352 Πέραν αυτών όμως, υπάρχουν και άλλες μορφές που δεν χρησιμοποιούνται παντού. Σε κάποιες περιπτώσεις επιτυχημένες, αλλά όχι σε όλες τις χώρες. Άλλη δυνατότητα λοιπόν ήταν να εναρμονίσουμε ε, την νομοθεσία για τη δημιουργία θηγατρικών και να περιορίσουμε τη δυνατότητα αυτή για τις ΜΜΕ. Αυτό θα ήταν όμως πολύ περιοριστικό. Πάλι θα ήταν δύσκολο να διαπραγματευτεί, να διαπραγματευτεί κανείς. Και γιατί να περιοριστούμε στις θηγατρικές μόνο, αφού το 98% όλων των εταιριών είναι ΜΜΕ, θα ωφελούνταν ούτως ή άλλως. Και αν άλλε εταιρείε πιο μεγάλε μπορούν να αποφεληθούν από την απλούστευση, γιατί να μην καλύψει και αυτές αυτό το μέτρο. Τρίτη επιλογή. Εναρμόνιση σε σχέση με τη θέσπιση θεατρικών υπό τη μορφή εταιριών δημόσιων και ιδιωτικών περιορισμένης ευθύνης. Μιλήσαμε με τα κράτη-μέλη πριν δρομολογήσουμε την πρόταση και με τους μπλεκόμενους φορείς και αυτή η επιλογή φάνηκε εξαιρετικά δύσκολη. Λόγω των παραδόσεων και δυσκολιών. Είναι δύσκολο να έχουμε ένα και μόνο μοντέλο στην Ευρώπη, το οποίο να αντικαταστήσει όλα τα εφιστάμενα. Υπήρχε επιλογή του να μην κάνουμε τίποτα. Πάλι θα ήταν δαπανηρό όμω να μετακατασταθούν στο εξωτερικό ε, κάποιε επιχειρήσει, γιατί θα έχουν να αντιμετωπίσουν 28 διαφορετικά εταιρικά δίκαια. Βάλαμε λοιπόν όλα αυτά, ε, τα είχαμε υπόψη μας, τα βάλαμε κάτω για να δούμε αν μπορούμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση που όμως να σέβεται ταυτόχρονα και τις εθνικές νομοθεσίες και να αντιμετωπίζει μόνο ακριβώς αυτά τα σημαντικά στοιχεία για το διασυναριακό εμπόριο για την ε, δημιουργία θεατρικών. Και έτσι καταλήξαμε στην έννοια της μονοπρόσωπης εταιρείας περισμένης ευθύνης. Ίσως είναι καλύτερη δυνατή προσφορά, μπορούμε να κάνουμε από τις παρούσες συνθήκες. Δεν μπορούσαμε να μην κάνουμε τίποτα, δεν ήταν επιλογή αυτό, γιατί οι πολίτες αυτό που περιμένουν από εμάς είναι να διευκολύνουμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη τη σύσταση συγκρότηση νέων εταιριών. Φυσικά δεν θέλω να πω ότι η πρόταση αυτή ομόνια της θα δημιουργήσει θέσει εργασίας. Πρέπει να είναι κατάλληλε και μακροοικονομικές συνθήκες και να υπάρξουν και πολλές άλλες μεταρρυθμίσει. Αυτό είναι ένα λιθαράκι. Σημαντικό λιθαράκι όμως. Μπορεί να συνεισφέρει στη διευκόλυνση τη δημιουργία, τη σύσταση επιχειρήσεων. Άρα, και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασία. Τι είναι αυτό το SUP όμω. Είναι συμβιβασμό μεταξύ μια εθνική και μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Ζητήσαμε λοιπόν από τα κράτη-μέλη στα εθνικά νομικά του συστήματα να προβλέψουν αυτή τη μορφή εταιρεία που θα είναι εθνική αλλά θα έχει κάποιε αναρμονισμένε απαιτήσει, άρα και μια κοινή ονομασία. Κάναμε διαβουλεύσει αυτή ήταν και η προτιμητή επιλογή. Το 57% των εμπλεκόμενων φορών συμφώνησαν. Και συγκεκριμένα επιχειρήσεις και οι ομοσπονδίες επιχειρήσεων συμφώνησαν. Αυτές δηλαδή ακριβώς που δημιουργούν αυτές τις εταιρείε, μπορούν να δημιουργήσουν αυτή τη μορφή εταιρεία. Στόχος της πρότασης λοιπόν είναι να ενθαρρύνουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα, να διευκολύνουμε τις διασυνορικές συναλλαγές, να αυξήσουμε τις διασυνορικές επενδύσεις, να προσαρμοστούμε στην ψηφιακή εποχή, οπότε στο τέλος να ε, αξιοποιήσουμε τον εκμετάλλευτο ακόμη δυναμικό ξένες αγορές. Τι ε, ε, τι προσφέρει αυτή η πρόταση, πρώτα απ' όλα. Κανόνες για αύξηση των διασυνορικών δραστηριοτήτων. Έχοντα υπόψη και την αναλογικότητα, δεν τα εναρμονίζουμε όλα και ούτε αντικαθιστούμε τους υφιστάμενους κανόνες. Απλά ζητάμε από τα κράτη-μέλη να προβλέψουν αυτό το ενδεχόμενο, αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή να μπορούν οι ιδρυτέ μια εταιρείας να, ε, να καταφύγουν σε αυτή την επιλογή. Και αν καταφύγουν σε αυτή την επιλογή, να υπάρχει αυτή η μορφή εταιρεία με το ενιαίο καταστατικό, με την κοινή ονομασία να μπορεί να ε, γίνεται η σύσταση εταιρεία ηλεκτρονικά, να υπάρχει αυτό το ελάχιστο κεφάλαιο κτλ. Άρα, ανταποκρινόμαστε στην αίτηση αυτή στο αίτημα του μανιφέστο, δηλαδή να μπορεί να υπάρχει ευκολία στη δημιουργία ε, και τη λειτουργία ε, μιας επιχείρησης δεσνοριακά. Άρα μια επιλογή προσφέρουμε. Και αυτό μας αρέσει τόσο πολύ. Είναι η επιλογή που προσφέρουμε στα κράτη-μέλη. Αυτά θα διαλέξουν πώς θα εφαρμόσουν αυτή την επιλογή. Αλλά θα έχουν ε, απλά προσθέσει μια νέα μορφή εταιρεία. Και θα το αφήσουν στους επιχειρηματίες να επιλέξουν αν θα επιλέξουν αυτή τη μορφή εταιρεία ή όχι. Αν δεν θέλουν μπορούν να επιλέξουν τις εθνικές μορφές εταιρεών. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι αν θέλουν κάποιες εταιρείε να αναπτυχθούν διασυνοριακά, το να έχουν αντιμετωπίσει 28 διαφορετικές νομοθεσίες δεν είναι και τόσο απλό. Ίσως λοιπόν τείνουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη νέα μορφή εταιρεία. Βλέπετε λοιπόν μια τυπική μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία εδρύεται σε μια, χώρα και αναζητεί επιχειρηματικέ ευκαιρίες σε μια άλλη. Φυσικά και μπορεί να παράσχει υπηρεσίες διασυνοριακά και ε, να ασχοληθεί με το διασυνοριακό εμπόριο. Θα πρέπει όμως να δημιουργήσει μια θηγατρική Πού αυτή η θεατρική θα είναι λοιπόν, λέμε τώρα μια SUP. Είναι ευκαιρία ή είναι κίνδυνος. Ήδη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην ακρόαση που έγινε στην Επιτροπή Γιούρη, με ακούσει κάποια σχόλια και είχα πει και εγώ κάποια σχόλια. Και ουσιαστικά διαρωτώ με κι εγώ ίδιος αν κριτική που άκουσα ε, οι επικρίσεις που άκουσα σχετίζονται όχι με αυτή την πρόταση. Διότι πολλά υπόθηκαν για την πρόταση αυτή. Ότι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο θα βοηθήσει στην ε, αύξηση των εικονικών εταιριών, αυτών των λεγόμενων εταιριών γραμματοκιβωτίου δεν θα προσφέρει επαρκή προστασία στους ε, πιστωτές, δεν θα σέβεται την νομοθεσία κατά του ξεπλήματος χρήματος. Περί του αντιθέτου πρόκειται όμως, διότι ακριβώς με το χρονοπλαίσιο προσφέρονται πιο πολλές δυνατότητε για ξέπλυμα χρήματο. Αντίθετα, εμεί θα προσφέρουμε αυτή την εταιρεία και λιγότερε δυνατότητε και θα προστατεύσουμε περισσότερο του πιστωτέ. Έχουμε τη διαδικασία τη δήλωση φερεγγιότητας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν διανέμονται τα μερίσματα και το καθεξής. Άρα φαίνεται να υπάρχει κάποια παρανόηση σε σχέση με αυτή την πρόταση και τις ευκαιρίες που προσφέρει. Εμείς πιστεύουμε ότι ο στόχος μας είναι και αυτό που θα πετύχουμε είναι ο εξυγχρονισμός. Απλούστευση απαιτήσεων, μείωση του ελάχιστου κεφαλαίου, ηλεκτρονική εγγραφή. Υπάρχουν αυτά ήδη. Δεν είναι ιδέες κομισιών. Είμαστε φιλόδοξοι μεν, αλλά κάποια κράτη-μέλη τα έχουν ήδη αυτά που σας προανέφερα. Έχουν ήδη ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι. Δεν το ελάχιστο κεφάλαιο στην Ευρώπη, θα δείτε την τάση. Υπάρχουν κράτη που πιστεύουν ακόμα ότι με το ελάχιστο κεφάλαιο προστατεύουν καλύτερα τους πιστωτές από την ασχοληθούμε με τα θέματα ρευστότητα και φερεγγιότητα. Αλλά αν εμβαθύνει κανείς στο ζήτημα του ελάχιστου κεφαλαίου και του ποιο είναι ο στόχο του τελικά, οι περισσότεροι βλεκόμενοι φορεί συμφωνούν ότι πιο πολύ είναι ένα κατόφλι για τη φήμη παρά προστασία των πιστωτών. Γιατί είναι στα βιβλία αυτό το ελάχιστο κεφάλαιο. Δεν σημαίνει ότι είναι και διαθέσιμο ως ρευστότητα, βλέπετε τώρα τα άλλα θέματα της επιγραμμικής ηλεκτρονικής εγγραφής. Υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη να της ηλεκτρονικής εγγραφής μιας εταιρεία και μια ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων στα μητρώα. Υπάρχουν βέβαια μεσάζονται σε κάποια κράτη-μέλη, σίγουρα, σε 16 όμως κράτη-μέλη ήδη υπάρχει απευθεία, ηλεκτρονική εγγραφή από τον ιδρύτη τη εταιρεία κατευθείαν στο Μητρό. Εξαιρέσει υπάρχουν, αλλά και εδώ υπάρχει η δυνατότητα εγγραφή από το συμβολογράφιο το μεσάζοντα στο Μητρό. Το σύστημα όμως υπάρχει ήδη. Ποια είναι η πρόταση. Τι θέλουμε να πούμε για την ηλεκτρονική εγγραφή. Θέλουμε να είναι βέβαιο ότι ο υπηρετής μπορεί διασυνοριακά, από απόσταση δηλαδή, και βέβαια με όλους τους δέοντες ελέγχους ε, πρέπει να γίνουν από το κράτος εγγραφής, καταχώρησης, που να απαιτήσει δηλαδή αυτό το κράτος διαδικασία εθνικών διασυνοριακών ελέγχων. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως είναι να υπάρχει η ηλεκτρονική εγγραφή καταχώρηση. Το πώς θα γίνει ακριβώς θα οργανώνεται από τα κράτη-μέλη μεμονωμένα. Δεν εντάσσεται στην πρόταση. Η υποχρέωση που υπάρχει είναι να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Ο τρόπος να πάει στα κράτη-μέλη. Ένα άλλο συχνό θέμα είναι αν υπάρχει διάκριση της έδρας κεντρικής διοίκησης από την έδρα της κύριας εγκατάστασης ή τον τόπο της κύριας εγκατάστασης. Πάντοτε προτείναμε Ε, ότι ναι, μπορεί να είναι διαφορετικές αυτές οι έντρε, άρα είμαστε συνεπεί στην πολιτική που έχουμε ακολουθήσει εδώ και κάποια χρόνια. Μπορούμε να δούμε αν αυτό θα μπορούσαμε να το διαπραγματευτούμε ή να το εξετάσουμε. Πιο προσεκτικά είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Όμω θέλω να σα υπενθυμίσω ότι για τι ερχόμενε εταιρείε ήδη υπάρχει νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Οι εταιρείε δηλαδή που έχουν ε, αλλού τα, την καταστατική τους έδρα από την ε, έδρα της κύριας δραστηριότητα. Σε κάποιες χώρες είναι, δυνατή, είναι δυνατός ο διαχωρισμός, όπως γίνεται και στη Γερμανία. Συμμετοχή τώρα των εργαζομένων. Θέμα εθνικού δικαίου. Και το αφήνουμε στην αρμοδιότητα, γιατί όπως είπα θέλουμε να εστιάσουμε μόνο στα στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για τη δημιουργία θηγατρικών στο εξωτερικό. Δεν κάνουμε μια πρόταση για τη μεταφορά καταστατικών ε, εδρών. Επέκταση είναι πιο πολύ, όχι κινητικότητα. Αν δεν υπάρχει κινητικότητα, δεν χρειάζεται ανάγκη να ρυθμιστούν αυτά τα ζητήματα, μπορεί να ρυθμιστούν στο εθνικό δίκαιο αλλά είμαστε ανοιχτοί σε συστάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά. Τώρα, Πασχόληση, εταιρείε, εικονικέ γραμματοκιβωτίο, τα είπαμε αυτά. Κατά την άποψή μας το εταιρικό δίκαιο δεν είναι και το πιο χρήσιμο εργαλείο για να δούμε αν υπάρχει ε, κατάχρηση του εργασιακού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά και δεν θα ήθελε να έχουμε εξαναγκαστική, καταναγκαστική αυτοαπασχόληση. Στηρίζουμε απόλυτα τον αγώνα κατά αυτών που εξαναγκάζουν κάποιον να γίνει αυτοαπασχολούμενος κατά κάποιο τρόπο. Είναι ένα φαινόμενο γνωστό και δεν μιλάμε στρικτό, στρικτό σένσου ε, για, για το τερικό δίκαιο. Πολλέ από τι εταιρείε αυτέ δεν είναι σε ευθύνη. Είναι εταιρείε περιόριστη ευθύνη, θα έλεγα, που δεν εμπίπτουν καν στο πλαίσιο μιας SUP. Πρόβλημα όμως υπάρχει με αυτή την λεγόμενη εξαναγκαστική αυτοαπασχόληση. Και θέλουμε να το καταπολεμήσουμε. Δεν υπάρχουν όμως στοιχεία που να αποδεικνύουν ή να δείχνουν ότι στις χώρες που υπάρχει το ελάχιστο κεφάλαιο, η ηλεκτρονική εγγραφή, έχουμε υψηλότερο ποσοστά αυτού του φαινομένου από αυτά που έχουν υψηλότερα, από τις χώρες που έχουν υψηλότερα κατόφλια και προϋποθέσεις για τη σύσταση εταιριών. Ευχαριστώ. Μίτσι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μίτσι. Καλημέρα σας. Πολύ ενδιαφέρουσα άσκηση ήταν αυτή, πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια και η δική μου προσέγγιση ήταν και είναι πολύ ανοιχτόμυαλη. διότι μετά από ενδελεχή εξέταση της πρότασης αυτής έχουμε εντοπίσει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και δίκαιοι και να διασφαλίσουμε ότι πραγματικά θα συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη της οικονομίας και πρέπει να είμαστε ανοιχτό μυαλί για να το κάνουμε αυτό. Εκτιμώ λοιπόν ότι το πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρησιμοποίησε, ε, Επιτροπής ε, χρησιμοποίησε αυτή την προσέγγιση. Οι μικρομεσαίες εταιρείες πολλές φορές αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες όταν θέλουν να επεκταθούν πέρα από τα σύνορα. Και τα προβλήματα, τα διασυνοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν έχουν να κάνουν με έξοδα, με νομοθεσία, με ρυθμίσεις και ε, όλα αυτά πολλές φορές εμποδίζουν τις εταιρείες από το να επεκταθούν, από το να μεγαλώσουν. Γι' αυτό λοιπόν Εκτιμώ πάρα πολύ το σκοπό αυτής της ε, πρότασης. Φυσικά και θέλουμε να διευκολύνουμε τις διασυνοριακές δραστηριότητες, διότι αυτό θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και την ανταγωνιστικότητα και αυτό θα γίνει προς όφελος των καταναλωτών εν τέλει. Και πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι το δυναμικό της ενίας αγοράς παραμένει ανεκμετάλλευτο. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε αυτό το δυναμικό πρώτα έτσι ώστε να μπορέσουμε να το εκμεταλλευτούμε έπειτα. Και μικρές λοιπόν εταιρείε, επιχειρηματίε που θέλουν να επεκταθούν βλέπουν ότι υπάρχει ένας μεγάλος κατακαιρματισμός της ψηφιακής ενίας αγοράς και αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε καλύτερα. Πιστεύω πως αυτή η πρόταση ενισχύει το επιχειρηματικό πνεύμα, κάτι που είναι αναγκαίο για την περαιτέρω εξέλιξη. Και την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο ο πρόεδρος ο Γιούνκερ μας παρουσίασε τις προτάσεις του και η ψηφιακή καινοτομία αποτελεί έναν από τον πυρήνα ε, και έναν από τους ε, πυλώνες αυτής της πρότασης. Ωστόσο, Δεν είμαι πεπισμένη ότι αυτή η πρόταση έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή αποτελεί λύση. Και για τους λόγους για τους οποίους ανέφερα. δεν μπορούμε να ενεργήσουμε εις βάρος των καταναλωτών, των εργαζόμενων και των δικαιωμάτων των πιστωτών όταν θέλουμε να επεκτείνουμε τις δυνατότητες μιας εταιρείας. Και πραγματικά πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα δικαιώματα των πιστωτών. Και μάλιστα υπήρξε μια διαφάνεια όπου μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι 50% των ενδιαφερομένων είναι υπέρ. Όμως ποιοι είναι αυτοί. Έχουν, έχουν ε, έχουν μπορέσει να πούν τη γνώμη τους τα συνδικάτα, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οργανώσει των καταναλωτών. Συνοψίζοντας λοιπόν θα ήθελα να πω ότι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η πρόταση και το λέω αυτό γιατί δεν μπορούμε να ενεργήσουμε βάση της πρότασης αυτής είναι ένα δημοσιονομικό όραμα το οποίο θα υπονομεύσει τα δικαιώματα των εργαζομένων της εταιρικής διακυβέρνησης Βέβαια θα μου πείτε ότι δεν χρειάζεται αυτή η πρόταση για να υπονομευτούν τα δικαιώματα. Όμως γιατί να δώσουμε και νέο, νέους τρόπους για να υπονομευτούν αυτά τα δικαιώματα. Το αντίθετο πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να δώσουμε ακόμα περισσότερες δυνατότητες για φοροαποφυγή. με το να δώσουμε την ευκαιρία στις εταιρείε να αναζητήσουν κάποιο καλύτερο καθεστώς αλλού. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή η πρόταση δεν περιορίζεται στις μικρομεσαίες εταιρείε. Μπορεί αυτό να ακούμε συνέχεια, όμως δεν περιορίζεται εκεί. Είναι διαθέσιμη σε όλες τις εταιρείε και στις πολυεθνικές ακόμα. Και δεν νομίζω πως οι πολυεθνικές έχουν ανάγκη αυτήν την νομοθεσία για να ε, δουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες που έχουν. Και δεν λέω πως αυτό είναι λάθος, απλά λέω πως υπάρχουν αρκετές δυνατότητες ήδη για τις πολυεθνικές ή για τις μεγάλες εταιρείες που θα τις διευκολύνουν να χρησιμοποιήσουν τη διασυνοριακή νομοθεσία. Δεν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για το ότι η δημιουργία αυτής της SUP θα αυξήσει τις διασυνοριακές δραστηριότητες, εμπορικές διαστηριότητε. Μια εταιρεία που θέλει να επεκταθεί διασυνοριακά έχει στη διάθεσή της ε, διάφορους κανονισμού. Εντάξει, υπάρχουν σίγουρα έξοδα, όμως πιστεύω πως όταν κάποιο θέλει να επεκταθεί σε κάποια άλλη χώρα, το έχει σκεφτεί στο βαρά το θέμα. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι η δημιουργία αυτής της ε, SUP θα αυξήσει τις δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκαν αυτά τα 230 έως 360 εκατομμύρια το χρόνο που θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποια απόδειξη γι' αυτό, δεν υπάρχουν δεδομένα γι' αυτό. Και Κάτι άλλο που είναι αμφιλεγόμενο έχει να κάνει με την ε, διοικητική έδρα μία εταιρεία και την καταστατική έδρα μία εταιρεία. Και αυτό πραγματικά μπορεί να δώσει αφορμές ε, για κατάχρηση. Βέβαια σίγουρα όλοι οι νόμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με καλό ή άσχημο τρόπο. Αλλά τέλος πάντων, κάτι άλλο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι αυτό το ελάχιστο κεφάλαιο του, ε, ε, του ευρώ. Όταν εμεί θέλουμε να εισαγάγουμε ένα νέο μέσο, και αυτό το λέω έχοντας υπόψη αρκετού που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, Πιστεύω πως, εντάξει, μπορεί να είναι συμβολικό ποσό το 1 ευρώ, όμως θα βρούμε μεγάλη αντίσταση μπροστά μας, διότι αυτό το συμβολικό ποσό του 1 ευρώ εξευτελίζει το, το σκοπό της νομοθεσίας. Οποιοςδήποτε σοβαρός επιχειρηματίας δεν ε, θα... Το, δεν θα προχωρήσει στη σύσταση μιας εταιρεία στο εξωτερικό επειδή θα τον τραβήξει αυτό το χαμηλό ποσό του ενό ευρώ. Εντάξει, σίγουρα διευκολύνει την εγγραφή μιας εταιρείας σε καταστατικό του εξωτερικού, όμως πιστεύω πως δεν εξυπηρετεί το σκοπό Χρειαζόμαστε επίσης ένα μητρό καταχώρησης μιας εταιρείας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι μια μικρομεσαία εταιρεία, ένας επιχειρηματίας φυσικά έχει να αντιμετωπίσει 28 διαφορετικές νομοθεσίες και ενδεχομένως 28 διαφορετικά έντυπα για να συμπληρώσει. Σίγουρα λοιπόν χρειάζεται κάποια ενιαία ρύθμιση. Όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θεωρώ πως πρέπει να βρούμε μία λύση προτού εμφανιστούν τα πραγματικά προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε τι εμποδίζει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, του επιχειρηματικού πνεύματος που τόσο μας λείπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι όπως λέτε. Και μάλιστα σε αντίθεση με την ασιατική επιχειρηματικότητα, με το αμερικανικό επιχειρηματικό πνεύμα και να δούμε πραγματικά εάν όντως θα αποτελέσει λύση αυτή η δημιουργία μιας SUP ή αν απλά θα οδηγήσει σε ακόμα περισσότερη κατάχρηση του υφιστάμενου συστήματος. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριο Στέφανιτς, σκιώδης ηγητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω πως υπάρχει ανάγκη απλοποίησης της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πως πραγματικά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της ενίας αγοράς. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως η δημιουργία αυτής της ε, μονοπρόσωπης ευρωπαϊκής εταιρείας είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, τουλάχιστον από πλευράς τυποποίησης. Εγώ πρέπει να πω ότι βλέπω μόνο θετικά πράγματα σε, αυτό εδώ το, σε αυτήν εδώ την πρόταση. Όσον αφορά το αρχικό κεφάλαιο του 1 ευρώ, πιστεύω πως αυτό θα είναι πλεονέκτημα μόνο για τις νεοσύστατες εταιρείε. Χρειάζεται να τονώσουμε την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και πρέπει να απλοποιήσουμε τα διοικητικά. Διότι αν ρωτήσουμε τους επιχειρηματίες για το ποιο είναι το σημαντικότερο εμπόδιο που τους ε, εμποδίζει να επεκταθούν θα μας πούν ότι είναι αυτή η γραφειοκρατία. Και πιστεύω πως πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτή τη γραφειοκρατία, γι' αυτό και η πρόταση αυτή θεωρώ πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Επίσης, πιστεύω πως χρειάζεται να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ανακμετάλλευτο δυναμικό της ενίας αγοράς. Και αυτή η πρόταση είναι μία από τις λίγες που προσπαθούν να σπάσουν τους ε, φραγμούς αυτής της ενιαίας αγοράς. Χρειάζονται μεν όμοια πρότυπα στην ενιαία αγορά, όμως δεν πιστεύω πως χρειάζεται και όμοια φορολογία. Πρέπει φυσικά να προσπαθήσουμε να τυποποιήσουμε, αλλά να τυποποιήσουμε τη διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως ε, έχει υποβληθεί αυτή η πρόταση για τη SUP. Αυτός είναι ο σκοπός της. Μία ανησυχία μόνο έχω και αυτή είναι η ηλεκτρονική εγγραφή. Ξέρω πως υπάρχουν πολλές χώρες που ήδη παρέχουν αυτή τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής, όμως κάθε χώρα έχει διαφορετική, διαφορετική διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το χρόνο και για το κόστος εγγραφής μιας νέας επιχείρησης στην πρόταση αυτή. Και αν η πρόταση αυτή σκοπεύει να τυποποιήσει αυτές τις διαδικασίες για την εγγραφή νέων εταιριών. Ευχαριστώ. Τόνι, έχεις το λόγο. Πραγματικά ακούγοντας ε, τους ε, σοσιαλιστές με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό. Ιδιαίτερα όταν αναφέρθηκαν στα συνδικάτα. Φυσικά και χρειάζεται απελευθέρωση, χρειάζεται μια ελεύθερη νέα Ευρώπη. Και οι εργαζόμενοι θα έχουν τα καλύτερα δικαιώματα όταν θα λειτουργεί και σωστά το σύστημα και ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα. Είναι λοιπόν μια καλή προσπάθεια προσπαθούμε να προχωρήσουμε. Η ηλεκτρονική εγγραφή είναι κάτι το πολύ ωραίο. Η Εστονία έχει μάλιστα και ηλεκτρονική ηθαγένεια, δηλαδή έχει προχωρήσει πάρα πολύ όσον αφορά την ψηφιοποίηση. Είναι μια χώρα ελεύθερη και αισιόδοξοι και φυσικά ναι, είναι καλό να έχουν τη δυνατότητα οι νέοι να ανοίξουν μια εταιρεία με ένα ευρώ. Δεν θέλουμε γραφειοκρατία ούτε να ε, φοβήσουμε τους νέους. Πρέπει να αλλάξουν οι εταιρείε και πρέπει να αλλάξει και ο κόσμος διότι δεν πάνε καλά οι μεγάλες βιομηχανίες στην Ευρώπη. Η Apple και η Google πάνε καλά. Το διαδικτυακό πάει καλά. Δεν πάει καλά ο άνθρακας. Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται με αυτές τις δύο εταιρείες, τις μεγαλύτερες εταιρείες, την Apple και την Google. Είναι εταιρείες που αξίζουν δισεκατομμύρια δολάρια. Γιατί λοιπόν έχουμε δισταγμούς γιατί δεν προσπαθούμε να γίνουμε σαν και αυτούς. Λιγότερες ρυθμίσεις, ευκολότερη πρόσβαση. Αυτό θέλω και γι' αυτό θα πολεμήσω. Εντάξει, λοιπόν. Γρήγορα, γρήγορα να δούμε λοιπόν ε, την άποψή μας. Ε, είναι σημαντικό η ζωή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να γίνει πιο εύκολη και ιδιαίτερα σε τόσο δύσκολες οικονομικές περιστάσεις όπως αυτές που διανύουμε οι άτομα τα οποία μπορεί να βρίσκονται χωρίς δουλειά, χωρίς απασχόληση και θέλουν να φτιάξουν μια δικιά τους εταιρεία να μην αναμπούν στην μαύρο παραοικονομία κτλ. Θέλουν να ξεκινήσουν κάτι, ένα εμπόριο ή να προσφέρουν υπηρεσίες και θέλουμε λοιπόν αυτό να γίνει εύκολα. Γι' αυτό ακριβώς και Ακριβώς ε, σε κάποιες υφέσεις μπορούμε να δούμε ε, τις νέες και νοτόμες επιχειρήσεις ε, να οδηγούν την επιστροφή στην ανάπτυξη. Αυτό διαφέρει από μια πολυεθνική που φτιάχνει ένα σωρό διάφορες μικρές εταιρείες, κάλυψη για να αποφύγει Συμφωνώ, δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε όμως οι μικρές επιχειρήσεις να μπορούν γρήγορα και αποτελεσματικά να μπορούν να ε, στηθούν και να αναγνωρίζονται στην αγορά. Ξέρω από την εργασία της Κομισιόν ότι πολλές χώρες ήδη έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό online. Ε, υπάρχει και εκείνο το τήσιο η ε, ετήσια απόδοξη, ε, δηλαδή όταν είναι περιορισμένη σε ευθύνη η εταιρεία ε, υπάρχει το θετικό ότι δεν μπορεί να σου πάρει κανείς το σπίτι και αυτό είναι πολύ θετικό για όσους το προσπαθούν αυτό. Η Κομισιόν έχει εξετάσει στην μελέτη αντικτύπου τι θα συνέβαινε αν αυτό αυξανόταν αντί για ένα ήταν 100.000, 1.000, 35.000 γιατί εγώ θα ήθελα να γίνει όσο γίνεται πιο εύκολο. Να κατανοήσουμε τους κινδύνους, να κατανοήσουμε ότι δεν θέλουμε κατάχρηση, αλλά θέλουμε να είναι εύκολο. Μήπως τυχόν δηλαδή ε, το φτιάξουμε περίπλοκο με κάθε πρακτική που ακολουθείται σε κάθε χώρα και τελικά ε, δυσκολέψουν τα πράγματα, δυσχερανθούν αντί να διευκολυνθούν. Θέλουμε πραγματικά εμείς να το καταστήσουμε πιο εύκολο για τις επιχειρήσεις μας, να μην υπάρχουν καταχρήσεις, αλλά δεν θα πρέπει, όπως είπα, να γίνει εξαιρετικά περίπλοκο. και έπειτα Δεν φαίνεται να έχουμε σκιώδη για τους πράσινους. Α, η κυρία Σέντρα. Ναι. Εμείς δεν έχουμε ακόμα ορίσει κάποιον σκιώδη, αλλά ε, η συγγήτρια είπε σωστά ότι αν θέλουμε να αξιολογήσουμε τους δυνητικούς κινδύνους, τότε μια ομάδα όπως ε, τα εργατικά συνδικάτο, η ΜΚΟ θα πρέπει να δώσει την άποψή της και αυτό στο πλαίσιο της, του, της μελέτης αντικτύπου. Αν δεν έχει γίνει μπορούμε να το κάνουμε στην Επιτροπή. Επίσης να τονίσω ότι βεβαίως το μέσο της επιγραμμικής ε, ε, εγγραφής είναι θετικό αν ο στόχος είναι η ευκολότερη ε, ε, εγγραφή, αλλά αυτό που είδαμε στην Εστονία δεν είναι μια ηλεκτρονική ηθαγένεια, δηλαδή ότι μπορεί κανείς να γίνει επιγραμμικά πολίτης της Εστονίας, απλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένας απλός τρόπος ταυτοποίησης ηλεκτρονική ε, δικαίωμα κατοικίας, δικαίωμα παραμονής. Πρέπει ωστόσο να εξετάσουμε τις δυνητικές επιπτώσεις για τη φορολόγηση και τα εργατικά δικαιώματα με διαβούλευση με τους εμπειρογνώμονες για να μην συμβουλευτούμε μόνο τις εταιρείε που μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέσα. Μασταλκά. Γκουε, δεν έχετε σχόλια, όχι, ακούτε, ωραία και δεν έχω σκιώδη EFTD. Η Εύελιν äh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την επεξεργασία αυτού του θέματος, γιατί σίγουρα δεν είναι καθόλου εύκολο θέμα. Και πραγματικά χρειαζόμαστε μια καλή ενιαία αγορά και για τις επιχειρήσεις και για τους ε, εργαζόμενους. Όμως πρέπει να προσέξουμε τα δικαιώματα που υπάρχουν στο εργατικό δίκαιο, στο δίκαιο των καταναλωτών. Ε, πρέπει να προσέξουμε αυτά τα δικαιώματα να μην κινδυνεύσουν, να μην διακυβευτούν. Και πραγματικά αυτή η πρόταση εδώ ε, περιέχει μεγάλους κινδύνους και πρέπει να εξεταστεί πάρα πάρα πολύ προσεκτικά. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν κάνει εκτιμήσεις αντικτύπου να είναι πραγματικές εκτιμήσεις αντικτύπου και όχι εκτιμήσεις από τις οποίες μπορεί να υποθέσει κανείς ότι δεν υπάρχει στην ουσία κάποια εκτίμηση αντικτύπου αλλά μια επιχειρηματολογία υπέρ της πρότασης της Επιτροπής. Ναι, και αυτό το θέμα με την ε, επιγραμμική εγγραφή πραγματικά ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, όμως δεν το βλέπω πουθενά στην εκτίμηση αντικτύπου. Δεν βλέπω πουθενά πώς θα χρησιμοποιηθούν, πώς θα εφαρμοστούν αυτές οι δυνατότητες επιγραμμικής εγγραφής όταν έχουμε 16 διαφορετικούς κανόνες ε, σε αντίστοιχα κράτη-μέλη. Και τι θα γίνει εάν πραγματικά δημιουργήσουμε εμπόδια με αυτή την προσπάθεια ρύθμισης. Δεν είναι επιχειρηματολογία σωστή αυτή που άκουσα και αυτό όχι μόνο ε, για την ηλεκτρονική εγγραφή αλλά και με το θέμα της ε, του κόστους του ενός ευρώ για την καταχώρηση μιας εταιρείας. Τι γίνεται, υπάρχει υποχρέωση ανάληψης ευθύνης σε κάποια κράτη, υπάρχει, υπάρχουν πολύ αυστηροτέρες προδιαγραφές σε κάποια άλλα κράτη-μέλη και αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν στην εκτίμηση αντικτύπου. Όμως δεν άκουσα τίποτα για αυτά. Και πραγματικά θέλω να μάθω εγώ τι σημαίνουν όλα αυτά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και για τους εργαζόμενους που θα δουλεύουν εκεί. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα που πρέπει να περιέχονται σε μια εκτίμηση αντικτύπου, διότι όταν ένα κράτος ζητά μόνο ένα ευρώ για την εγγραφή μιας εταιρείας, τότε αυτό σημαίνει ένα ευρώ οι ίδιες απαιτήσει για όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους. Τι γίνεται όμως τα υπόλοιπα με που έχουν διαφορετικές ρυθμίσεις, διαφορετικούς κανόνες. Μήπως θα ανοίξουμε το δρόμο σε ορισμένες εταιρείε έτσι ώστε αυτές να έχουν τη δυνατότητα να ε, καταχωριστούν σε μια άλλη χώρα χωρίς για παράδειγμα τη σύμφωνη γνώμη των ε, εργαζομένων τους όπως πρέπει να γίνεται στη Γερμανία. Και εδώ δεν μιλάω για μικρές επιχειρήσεις, μιλάω για μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν ένα με εξίσου μεγάλο νομικό επιτελείο που θα εκμεταλλευτεί κατάλληλα την κατάσταση. Πιστεύω πως πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να δούμε προτού προχωρήσουμε. Και εδώ πέρα συμφωνώ απόλυτα με την ε, κυρία Μίτση διότι πραγματικά έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας και πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για διευκρινήσεις. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει το κείμενο που έχουμε. Σχεδόν δεν έχουμε άλλο χρόνο, έχουμε τέσσερις ακόμα μελητές όμως και θα ήθελα και η Κομίσιον να μπορέσει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ σύντομα θα υπάρξει και άλλος γύρω συζήτηση το Φεβρουάριο έτσι κι αλλιώς για το θέμα αυτό όταν θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. Η Μαρία Γουαρτίνη και Κάφεν και Γιούρι. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω λοιπόν να χρησιμοποιήσω αυτό το ένα λεπτό για να πω αυτά που ήθελα να πω. Καταρχάς θα ήθελα να πω στους ε, συναδέλφους ότι Εγώ έχω εργαστεί 25 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, έχω ιδρύσει επιχειρήσεις και έχω επιφυλάξεις. Και θα σας πω γιατί έχω επιφυλάξεις, γι' αυτό ζήτησα το λόγο, γιατί υπάρχουν εμπόδια, υπάρχουν φραγμοί ακόμα και τώρα που δεν έχουμε αυτές τις ρυθμίσεις. Υπάρχουν, λοιπόν, και το ξέρω αυτό από τη Ρουμανία που έχω δραστηριοποιηθεί, πάρα πολλά εμπόδια τα οποία καθιστούν αδύνατη την επέκταση μιας εταιρείας. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν χάσει τη δουλειά τους εξαιτίας αυτών των εμποδίων. Υπάρχουν εταιρείες που συνεργάστηκαν με άλλες εταιρείες, αγοράστηκαν και μετά απολύθηκαν οι εργαζόμενοι. Πιστεύω πως ε, όταν έχουμε λοιπόν ένα ενιαίο έγγραφο, ένα ενιαίο ρυθμιστικό έγγραφο που θα χρησιμοποιείται και στα 28 κράτη-μέλη θα έχουμε ήδη κάνει πάρα πολλά προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως, ε, θα ήθελα να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτή δεν είναι μελέτη, αυτή είναι παροδία πραγματικά. Περί, είχαμε περίπου 500 απαντήσει από πάρα πάρα πολλούς ενδιαφερόμενους και φορεί. Αυτό πραγματικά δεν είναι εκτιμήση αντικτύπου και όταν κάνατε κάποιες εκτιμήσεις κινδύνου πρέπει να είναι μακροπρόθεσμες και όχι ε, βραχυπρόθεσμες. Πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί στις αναλύσεις μας διότι αυτό που θέλουμε είναι να βελτιώσουμε τα πράγματα, όχι το αντίθετο. Έτσι όμως όπω μα έχετε παρουσιάσει τα πράγματα δεν γίνεται αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ακούσει πράγματα που τα έχω ξαναπεί στην Επιτροπή Γιούρι. Θέλω όμως να τα επαναλάβω σε αυτήν την Επιτροπή. Καταρχάς, διατυπώσεις για την ηλεκτρονική καταχώρηση. Δεν υπάρχει μόνο η Εστονία, θα σας πω και για τη χώρα που ξέρω πολύ καλά, τη Γαλλία, τι γίνεται. Στο πλαίσιο της οδηγίας για τις ε, υπηρεσίες, η Γαλλία προβάλλεται ως μία από τις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις και επιλέξαμε στη Γαλλία τη δημιουργία όλων των επιχειρήσεων, ακόμη και αυτών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της οδικές για τις υπηρεσίες. Όλες οι επιχειρήσεις. Αν λοιπόν ο στόχος τελικά είναι όλες, σε όλα τα κράτη-μέλη να είναι δυνατόν όλες οι διατυπώσεις την δημιουργία επιχείρησης να γίνονται ηλεκτρονικά, είναι μια καλή πρόταση, έτσι. Θα ήταν αυτό μια πάρα πολύ χρήσιμη πρόοδος. Όμως, ερωτώ, πρέπει να γίνει εναρμόνιση εταιρικού δικαίου για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και γιατί είδους εναρμόνιση μιλάμε. Γιατί είδαμε κάποια κριτήρια που θα εφαρμόζονται για αυτή την Ευρωπαϊκή Μονοπρόσωπη Εταιρεία. Είναι μέγιστη εναρμόνιση αυτή, δηλαδή αυτού του είδους η εταιρεία θα ε, έχει αυτά τα κριτήρια όλα και μόνο αυτά τα κριτήρια και μόνο αυτή. Δεν καταργούνται όλες οι ασφαλιστικές δικλείδες που ήθελαν να δημιουργήσουν οι χώρες για την προστασία των πιστωτών και των μισθωτών. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Και η συγκήτρια είπε επίσης ε, πολλά. Ή μήπω τελικά είναι ένα ελάχιστη εναρμόνιση, δηλαδή ένας ελάχιστος κοινός παρονομαστής, οπότε τα κρατημέλη μπορούν να έχουν αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες που κρίνουν απαραίτητες για την προστασία πιστωτών, μισθωτών και να υπάρχει βέβαια ταυτόχρονα μια καλή ε, επικοινωνία με τις επιχειρήσεις και αντιστοίχησης. Έχουμε ήδη κάποιο είδους αντιστοίχηση χωρίς να είναι και κατηγορηματικά τα θετικά τα αποτελέσματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μονοπρόσωπες εταιρείε, βλέπουμε ότι πολλές φορές υπάρχει κατάχρηση του εργασιακού δικαίου με τη χρήση εταιριών σε τομείς που ξέρουμε πολύ καλά στην Επιτροπή αυτή όπως αυτή της οδηγίας για τις υπηρεσίες όπου συχνά βλέπουμε να έχουμε προσωρινή παροχή υπηρεσιών με πλαστούς ή εικονικούς αυτοαπασχολούμενους. Βέβαια, σίγουρα εδώ μιλάμε για αυτό. Απασχολούμαστε και όχι για τι μονοπρόσωπε εταιρείε περιορισμένη ευθύνη. Έχουμε όμω εντοπίσει τέτοια κρούσματα. Είναι ένα πραγματικό πρόβλημα και παρακάμπτεται η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων με την προσωρινή παροχή υπηρεσιών και με το καθεστώ των ψευδοαυτοαπασχολούμενων όπου ε, ε, και είναι δύσκολο να εντοπίσουμε την διάσταση του προβλήματος, επειδή είναι συγκαλυμμένα όλα αυτά και είναι δύσκολο να καταλάβει κανεί που είναι η κατάχρηση. Τώρα, η ευκολία πρόσβασης στη δημιουργία επιχείρησης επηρεάζει την εξαναγκαστική αυτοαπασχόληση. Το 24, ε, τη διαφάνεια 24, δεν ξέρω. Στη Γαλλία διευκολύναμε σημαντικά τις δηλώσεις για τους αυτοαπασχολούμενους και για θετικά αποτελέσματα μπορούσαν να ε, τακτοποιήσουν και να νομιμοποιήσουν τη δραστηριότητα που μέχρι τότε γινόταν ε, παρανόμως. Παράγματι όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι που εξαναγκάζονται να καταχωριστούν, να εργραφούν, ε, να είναι μισθωτοί. Η θα ήθελε να ασχοληθεί με τη δημιουργία επιχειρήσεων και ίσως έτσι τους δίνουμε ε, έναν ενθουσιασμό να το κάνω. Όμως, παρότι πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρα πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, θα πούμε στους νέους, ακούστε, μη συστήστε με πιέση, δηλωθείτε ως αυταπασχολούμενοι κτλ. Peut-être qu'on pourrait se lancer sur de la sans harmonisation sociale et sans harmonisation fiscale. Χωρίς φορολογική κοινωνική εναρμόση θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τα στρεβλά φαινόμενα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος, αφού είχε διακόψει την ομιλήτρια. Κοιτάξτε, προσπαθώ να παραμείνουμε στο χρόνο. Είναι σημαντικό το θέμα, αλλά έχουμε και άλλη συζήτηση που έχουμε προγραμματίσει. Η Κάθριν έχει τώρα το λόγο. Θα είναι πάρα πολύ σύντομα και το πρώτο κομμάτι της παρουσίασης. Είπατε 2% μόνο των ΜΜΕ επενδύουν στο εξωτερικό. Θέλω κάποιε περισσότερε πληροφορίε. Είναι παρόμοιε αυτέ οι επιχείρησει το 2%. Επίση, μελέτη αντικτύπου. Πολλοί ασχολούνται και κάποιε ομάδε έχουν αποκλειστεί από αυτή τη μελέτη αντικτύπου. Για το μέλλον είναι σημαντικό να έχουμε μια πιο έτσι ε, αντιπροσωπευτική μελέτη αντικτύπου. Επίσης, το ανθρώπινο κεφάλαιο έχει την αξία τους επιχειρήσει και θα πρέπει να διαφωνήσω με κάποια σχόλια ορισμένων συναδέλφων. Μπορεί να ανθεί η οικονομία, αλλά να έχουμε και κοινωνικά δικαιώματα, έτσι. Δεν πρέπει να το χάνουμε αυτό. Εσείς παρακαλώ. Πρόεδρε, έχω ένα σύντομο σχόλιο. Εγώ υποστηρίζω την πρόταση αυτή, αλλά άλλοι εξέφρασαν ανησυχία σε σχέση με το ελάχιστο κεφάλαιο του 1 ευρώ. Εγώ θέλω να στηρίξω αυτή την πρόταση. επειδή βόση εμπειρία που έχω από την Τσεχική Δημοκρατία, ε, ε, διατέλεσα υπουργό δικαιοσύνη και είχαμε μηδενικό ελάχιστο κεφάλαιο για τις εταιρείε και έτσι είδαμε αύξηση στην ε, δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Αν οι εταιρείε πρέπει να έχουν 100.000 ή 200.000, αυτό δεν σήμαινε απαραίτητα περισσότερη προστασία των πιστωτών. Αυτό που είδαμε ήταν ε, ε, ψευδή ελάχιστα κεφάλαια και οι επιτυχείς επιχειρηματίες είχαν συνήθως περισσότερα προβλήματα στο να στήσουν τις εταιρείες τους. Ε, κατανοώ τις αμφιβολίες σας και τις ανησυχίες σας. Πάντως δεν σημαίνει το ψηλότερο ελάχιστο ποσό και μεγαλύτερη προστασία. Αν ε, θέλουμε να δούμε πώς θα προστατεύσουμε τους ε, επιχειρηματίες, θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους. Δύο προτάσεις τώρα έχει ο τελευταίος. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να στηρίξω εγώ τον προηγούμενο μιλητή. Είχαμε παρόμοιες περιστάσεις στην Πολωνία όπου η δημιουργία μιας μικρής εταιρείας με περιορισμένες ευθύνες απαιτούσε 50.000 λότι αρχικά ο κεφάλαιο, πάνω από 10.000 ευρώ. Πριν από, λίγες, ε, λίγα χρόνια μειώθηκε αυτό το μήνυμο κεφάλαιο στα 1200 ευρώ. Και ωστόσο Είναι κόστος το οποίο καταναλώνεται στη διάρκεια της, ε, της καταχώρησης της εταιρείας. Δεν υπάρχει μηχανισμός δηλαδή έτσι και αλλιώς εξασφάλισης των πιστωτών. Ή θα, είτε είναι ένα ευρώ το κατόφλι, είτε είναι 100.000 δεν έκανε διαφορά όσον αφορά την προστασία των πίστοτων. Ξέρω πως δεν έχουμε χρόνο. Μία σύντομη πρόταση να πω. Ναι. Εμείς έχουμε εισάγει τις αλλαγές το 2009 Έχουμε το μήνυμα αρχικού κεφαλαίου και δεν εμφανίστηκε καμία παθολογία και κανένα πρόβλημα εδώ και πέντε χρόνια που ισχύει αυτό. Δεν έχουμε διαπιστώσει άδικες πρακτικές στην αγορά. Απλά αποδεικνύεται ότι στη σύγχρονη οικονομία δεν εγγυάται το κεφάλαιο την ε, δραστηριότητα και τη λειτουργία. Ευχαριστώ και τώρα η Κομισιόν και πάλι. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατανοώ το χρονικό περιορισμό και θα είμαι σύντομο, αλλά θέλω να απαντήσω πληρέστερα για το ελάχιστο κεφάλαιο, αλλά κατά κάποιο τρόπο αυτό απαντήθηκε από τους επόμενους ομιλητές που έδωσαν ακριβώς ε, το ίδιο, την ίδια ανάλυση που και εγώ θα έδινα, γιατί ξεκίνησα λέγοντας ε, πως η πρόταση αυτή θα έπρεπε να αφήσει μια επιλογή και στους επιχειρηματίες, γιατί δεν πιστεύουμε το ότι ε, τα κράτη θα πρέπει να υπαγορεύουν πόσο κεφάλαιο θα πρέπει να έχει αρχικά, θα πρέπει να είναι 50.000, 25.000 ή 5.000. Αυτό είναι έτσι κι αλλιώς ένας αυθαίρετος αριθμός. Δεν πιστεύουμε στους αυθαίρετους αριθμούς, αλλά αντίθετα άλλοι είναι οι ε, παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις. Μπορεί να ξεκινήσει κανείς με ένα ευρώ, αλλά δεν χρειάζεται ε, να έχει παραπάνω. Σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα στη Γαλλία, ξεκινούν με περισσότερα χρήματα, ακόμα και αν επιτρέπεται να έχουν χαμηλότερα ποσό. δεν χρειάζεται να μπει κάποιο συγκεκριμένο όριο. Είναι πολύ σημαντικό για τις καινούριε εταιρείε αν μιλάμε για ρευστότητα, πρόσβαση στη χρηματοδότηση κτλ. Και λέμε μετά ότι μια εταιρεία καινούργια πρέπει να έχει 65.000 ευρώ μίνιμουμ ε, κεφάλαιο. Μα δεν είναι αυτό που βλέπουμε στην πράξη και αυτό που πραγματικά είναι προστασία των πιστωτών είναι τι, αυτό που υπάρχει εδώ σε αυτή την πρόταση. Φερεγγιότητα, να δούμε δηλαδή πόσα κονδύλια έχεις και αν δεν έχεις θα είσαι προσωπικά υπεύθυνο. Εδώ λοιπόν προβλέπεται μεγάλο κομμάτι προστασίας σε αυτή την οδηγία. Σύντομα για τρία άλλα θέματα. Μελέτη αξιολόγησης. 30 σελίδε είναι αυτή σύμφωνα με τις κατευθυντήριε μα γραμμέ. Πραγματικά, αν εσεί καταφέρετε να βάλετε όλε αυτέ τις πληροφορίε για όλα τα κρατημέλη, όλε τι εργατικέ νομοθεσίε και τι νομοθεσίε περί προστασίας των πιστωτών σε 30 ε, σελίδες, ε, θα σα χαρίσω ό,τι θέλετε. Έχουν γίνει πολλές αναλύσεις, σίγουρα όμως σε 30 σελίδες δεν μπορούμε να αναλύσουμε τα νομικά συστήματα των κατορμελών. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερα, αν πιστεύετε πως δεν είναι αρκετά, Μπορείτε να το συζητήσετε, αλλά σε σχέση με τε, τους διαφορετικούς κανόνες για την καταχώρηση των εταιριών. Ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Τώρα οι εταιρείε λειτουργούν, μπαίνουν στην εσωτερική αγορά, αναγνωρίζονται ως εταιρείε και άρα πρέπει να αναγνωρίζουμε αυτούς τους κανόνες. Συμφωνώ ότι μπορεί να υπάρχει δυσκολία όσον αφορά τη διασυνοριακή τους αναγνώριση και εδώ η Κομισιόν και μπορούσε να αναφερθεί σε ένα νέο κανονισμό, στον νέο κανονισμό που άρχισε πρόσφατα να ισχύει, ε, για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των εταιριών. Ίσως αυτό θα είναι ένας τρόπος να αναφερθούμε σε αυτόν τον κανονισμό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και ε, ως λύση. Τέλος, η διαβούλευση έγινε online, ε, όπως κάνουμε και με άλλες ε, διαβουλεύσεις. Είναι αλήθεια ότι αυτές οι διαβουλεύσεις για πολλούς λόγους είναι ανοιχτές για όλους και για τους επιχειρηματίες αλλά και για τα συνδικάτα, τα οποία συνδικάτα συμμετείχαν στην online διαβούλευση. Αλλά ε, εντάξει, δεν είναι ιδανικό το μέσο αυτό, γι' αυτό και προσβλέπουμε στη συνεργασία με όλους τους ε, ε, εμπλεκόμενους φορείς, εάν θεωρούν πως δεν αντιπροσωπεύτηκαν ακριβώς στη διαβούλευση. Πάντως, αυτό η online διαβούλευση μας δίνει μια γεύση για το τι συμβαίνει επί τόπου. Περισσότερη διαβούλευση λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει όντω να γίνει ε, ηλεκτρονικά. Η είναι. Γρήγορα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ, πολύ καρποφόρα η συζήτηση. Συμφωνούμε όλοι εδώ ότι Είμαστε υπέρ το να αυξηθούν οι επιχειρήσεις, αλλά δεν συμφωνούμε απόλυτα για το πώς θα γίνει αυτό. Πάντως η συζήτηση ε, επικεντρώθηκε στο κεφάλαιο του ενός ευρώ. Όμως αυτό είναι μόνο ένα μέτρο. Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ νομίζω πως θα πρέπει να συμφωνήσουμε για κάτι το οποίο όλοι συμφωνούμε. Δηλαδή, να βρούμε τον τρόπο ώστε να διευκολύνουμε με ασφαλή τρόπο τους πιστωτές, τους εργαζόμενους, τους επενδυτές να αυξήσουν τις, ε, ε, τις επιχειρήσεις εν γέννη. Γι' αυτό και υποστηρίζω. Να βρούμε τον τρόπο ώστε κανείς να μην ζημιωθεί και είμαι πρόθυμη να ακούσω σε κάθε πρόταση με ανοιχτό μυαλό ώστε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο να προχωρήσουμε και να ε, προωθήσουμε τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ και φαντάζομαι πως θα συντάξει την εκθεσή σου μέχρι 16 Δεκεμβρίου. Οπότε σε ευχαριστώ πολύ και για όλη τη δουλειά που κάνεις. Ελπίζουμε λοιπόν ότι έτσι θα διευκολύνουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στην αγορά. Και πάμε τώρα στην δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ε, για τη συνεργασία όσον αφορά την πρόληψη και την αποφυγή της μη δηλωμένης εργασίας. Ντένις Γιώμ από την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Πιστεύω πως η ότι Θα η εργασία είναι λίγο σαν τη διαφθορά. Όταν δηλαδή αρχίζει, είναι δύσκολο να μην την ακολουθήσουν και οι άλλες εταιρείε. Διότι έχουν κάποια ωφέλη φυσικά όταν πληρώνεις λιγότερο τους εργαζομένους σου. Και αυτά που λένε πολλοί εκπρόσωποι μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ότι δεν θέλουν να χρησιμοποιούν αδίλωτη εργασία, αναγκάζονται όμω να το κάνουν επειδή το κάνουν και ανταγωνιστέ. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενώσουμε τι δυνάμει μα και θα παρακαλούσα για λίγη ησυχία σε αυτό το σημείο. Να ενώσουμε λοιπόν τις δυνάμεις μας για να προσπαθήσουμε να το καταπολεμήσουμε. Πιστεύω πως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα ενώσει όλες αυτές τις ε, επιθεωρήσεις εργασίας είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Έχω κάποιες παρατηρήσεις για την πρόταση αυτή και θα είμαι σύντομος. Θα είμαι σύντομο, διότι πραγματικά με ενδιαφέρει αντίδραση τη Επιτροπή αυτό. Καταρχάς, δεδομένη της πολιτικής σημασίας της πρότασης, πιστεύω πως πρέπει πραγματικά να τονίσουμε ότι αυτό είναι μόνο ένα από πολλά μέτρα που μπορεί να λάβει κανείς για να καταπολεμήσει την αδήλωτη εργασία. Η δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα ε, φέρει κοντά τις ε, διάφορες επιθεωρήσεις εργασίας χωρίς να ε, λαμβάνει όμως υπόψη την νομοθεσία είναι κάτι ελλειπές. Θα ήθελα λοιπόν να μου δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιβεβαίωση του ότι αυτό το μέτρο είναι ένα μέτρο από μία δέσμη μέτρων καταπολέμησης του προβλήματος αυτού. Έπειτα, δεδομένη επίση τη σημασία του θέματο, πιστεύουμε πω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει άμεση ανάμειξη στο θέμα. Γι' αυτό λοιπόν και χρειάζεται ένα εκπρόσωπό του για να συμμετέχει σε αυτήν την πλατφόρμα. Επίσης, οι αιτήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπή για τον τρόπο λειτουργία αυτού του συστήματος είναι κάτι αναγκαίο. Και εδώ χρειάζεται η συμμετοχή, η ενεργό συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αν διαπιστώσουμε ότι δεν λειτουργεί όπω θα έπρεπε αυτό το σύστημα, τότε θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να επηρεάσουμε διαφορε αλλαγε Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πω αυτε οι αιτήσει εκθέσει δεν θα πρέπει να είναι θέμα ρουτίνα, αλλά πραγματικά να εξετάζουν κάτω από το μικροσκόπιο το πώ λειτουργεί. Έπειτα, πεδίο εφαρμογή. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει μεν την αδήλωτη εργασία και την ε, πλασματική αυτοαπασχόληση, αλλά όχι άλλες ε, μορφές. Υπάρχει για παράδειγμα... Ε, υπάρχουν για παράδειγμα εταιρείε που λένε ότι πληρώνουν τους εργαζόμενους τους περισσότερο από ό,τι όντως τους πληρώνουν ή που τους δηλώνουν λιγότερες ώρες από εκείνες που πραγματικά έχουν εργαστεί. Επίσης πιστεύω πως πρέπει να κοιτάξουμε και αυτές τις μορφές της για μένα λάθος δηλωμένη εργασία. Επίσης πιστεύω πως πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις επιχειρησιακές δραστηριότητες. Έχουν γίνει συναντήσεις εμπειρογνωμόνων και το θυμάμαι αυτό και από τη δεκαετία του 90 στα, στις εσωτερικές υποθέσεις στα θέματα δικαιοσύνη. Τα θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί. Ε, πιστεύω πω ωραία είναι, όμω δεν έχουμε χρόνο για κάτι τέτοιο και πω πραγματικά θα πρέπει να δώσουμε την προσοχή μα στο πώ μπορούμε να συνεργαστούμε, πώ μπορούν να συνεργαστούν αυτέ οι επιθεωρήσει εργασία. Και επίση σημαντικό είναι να γίνουν ενημερωτικέ εκστρατείε από τις ε, Βρυξέλλες, αλλά και όχι μόνο από τις Βρυξέλλες. Πιστεύω πως πρέπει να μας βοηθήσουν εδώ οι κοινωνικοί εταίροι και τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν το καθένα ξεχωριστά μια δική του ενημερωτική εκστρατεία. Επίσης, πιστεύω πως η συμπερίληψη των κοινωνικών εταίρων στην δημιουργία αυτής της πλατφόρμας τουλάχιστον έτσι όπως φαίνεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, περιορίζεται τις περιπτώσεις όπου οι κοινωνικοί εταίροι έχουν και κάποιο ρόλο στην εφαρμογή, στην επιβολή. Και κύρια τον των κοινωνικών εταίρων, όπω είπα, είναι να αποτρέψουν κάτι τέτοιο από το να συμβεί. Στην πράξη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και γι' αυτό πιστεύω ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει πάντα να συμπεριλαμβάνονται, τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο, στις προπαρασκευαστικές εργασίες αυτή τη πλατφόρμα. Αυτά από μένα κύριε Πρόεδρε και ανυπομονώ να ακούσω τι απόψει των υπολείπων. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω δύο-τρία σημεία. Πρώτα απ' όλα, Πράγματι πρέπει να καταπολεμήσουμε την αδήλωτη εργασία. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Ωστόσο πρέπει να πω ότι ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο είναι με τη σωστή κοινωνική και φορολογική πολιτική. Και αυτά είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεν θα πρέπει λοιπόν να, να τα υποκαταστήσουμε μετατοπίζοντας την αρμοδιότητα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό, διότι Μιλάμε για μια πλατφόρμα. Ίσως όμως τελικά γίνει μια ε, μετατόπιση και τελικά μεταφορά αρμοδιοτήτων. Αυτή η πλατφόρμα έχει στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. Αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο. Όμως η αρμοδιότητα των κρατών μελών στον τομέα αυτό είναι ξεκάθαρη και ελπίζω να μην ε, αλλάξει. Επίσης, διαπίστωσα ότι υπάρχει αιτιολογημένη γνώμη από τα κράτη-μέλη για την πλατφόρμα αυτή. Εκεί επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν αρκετές και σαφείς πληροφορίες για τη σχέση μεταξύ της λειτουργίας της πλατφόρμας και τη μείωση της αντίληψης εργασίας και εκφράζεται επίσης η ανησυχία για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ συγκεκριμένα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, η Μαρία, Μαρία Γκουαρτίνη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και μιλώ για τους συντρόφους μου από την ομάδα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών επειδή είμαι σκιώδης εισηγήτρια. Αλλά και τον κύριο Ντε Γιόγκ θέλω να ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε. Δοθήκαμε αρκετές φορές, συζητήσαμε και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είναι πράγματι αυτή η πλατφόρμα χρειάζεται. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το ότι συμφώνησε με τις προτάσεις της σοσιαλιστικής ομάδας και συγκεκριμένα για να έχουμε ετήσιες εκθέσεις και όχι κάθε τέσσερα χρόνια. Και δέχτηκε και την πρόταση ότι θα πρέπει να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι πεπισμένη ότι η εν λόγω πλατφόρμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε διασύνδεση όλων των χωρών. Και εδώ Θέλω να υπογραμμίσω το γεγονό ότι θα πρέπει να είναι δεσμευτικό, υποχρεωτικό, όχι να επιλέξουμε ποιε χώρες θα είναι εντός και ποιε θα μείνουν εκτός. Αν θέλουμε να διασυνδέσουμε στην πλατφόρμα αυτή τα κράτη-μέρη, μέλη, συγγνώμη, θα πρέπει και το κοινοβούλιο να συμμετέχει, να ορίσουμε ένα άτομο συγκεκριμένο. Και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συμμετέχουν. Έτσι Ίσως περιορίσουμε κατά ένα μέρος την αδειλωτή εργασία, δεν μπορούμε να την εξαλείψουμε εντελώς ως φαινόμενο, μπορούμε όμως να μετριάσουμε αυτό το φαινόμενο και επίσης να διδαχθούμε και από τις καλές πρακτικές άλλων χωρών. Ελπίζω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει με θετικό μάτι τις προτάσεις μας. Θα μεταφέρω και άλλες υποδείξεις στον εισηγητή. Υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις γλωσσικού χαρακτήρ. κάποια ε, μικρό αλλαγή στη διατύπωση θα προτείνω. Κατά τα λοιπά συμφωνούμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ξονόματος ομάδας ECR δεν είναι εδώ δυστυχώς ο Σκιώδης, αλλά μου έδωσε τις σημειώσεις του. Στηρίζει την αρχή της πλατφόρμας και την εστίαση σε δράση επιβολής. Επίσης, το σχόλιο που κάνατε κύριε Ντεγιόγκ για την καταπολέμηση της αδηλώτης εργασίας και της υποδηλωμένη εργασίας. Είμαστε σύμφωνοι ως προς την αρχή, αλλά το να είναι υποχρεωτική συμμετοχή είναι κάτι που μας προβληματίζει δεδομένων των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών. Παραλαμβάνουμε, έχουν τα κράτη-μέλη την αρμοδιότητα. Το είπε και το ΕΛΚΟ. Συμφωνούμε ότι πρέπει να είναι οικονομικά συγγνώμη, αποδοτικό για τα κράτη-μέλη. Φυσικά η αδηλωτή εργασία περιορίζει τα έσοδα. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη εντός της δικαιοδοσίας τους να προβούν στα μέτρα. για την γρήγορη αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφόρων συμφωνούμε όπως και εν γέννη συμφωνούμε με την ανταλλαγή δεδομένων, βέλτιστων πρακτικών. Αλλά υπάρχουν και βέστα ζητήματα όπως είναι οι αρχές της προστασίας δεδομένων που όταν μιλάμε για τα οικονομικά των ε, προσώπων. Αυτό πρέπει να το εντάξουμε σε μια ευρύτερη συζήτηση για την προστασία των δεδομένων. Επίση, η ανταλλαγή πληροφοριών γνωρίζουμε ότι μπορεί να είναι και ακρό δαπανηρή, άρα θα πρέπει να γίνει με αναλογικό τρόπο προ το επίπεδο τη παράβαση. Διότι αν υπόκειται για τη συνορική δραστηριότητα και γι' αυτό θα καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες. Τώρα ε, ε, για την ομάδα ALDE, κυρία Κάλλας. Ευχαριστώ. Εγώ εκπροσωπώ την ALDE, ξενόμα της κυρίας Τονάης, ε, και διαβάζω ένα έγγραφο το οποίο μου έδωσε. Ζητεί συγγνώμη που δεν μπορούσε να είναι παρούσα, αλλά είναι αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Απασχόλησης και θα παρακολουθήσει τη συζήτηση και στις δύο επιτροπές. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Εν γέννη στηρίζουμε την ιδέα μιας νέας πλατφόρμας, καθώς σημαίνει ε, επιθεωρητές εργασίες, σε φορολογικές αρχές καθώς και, κοινωνικές αρχές, ε, και κοινωνικούς εταίρους. Είμαστε πεπισμένοι πως η ανταλλαγή ε, βέλτιστων πρακτικών θα βελτιώσει την κατάσταση των μη διδηλωμένων εργαζομένων, θα διευκολύνει τη συνεργασία και θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να μάθουν τι συμβαίνει, όμως θα πρέπει να καλύψουμε αυτά που, ε, να, μάλλον, να μην ε, υπερκαλύψουμε αυτά που ήδη υπάρχουν, αλλά και να σεβαστούμε τα μοντέλα της εσωτερικής αγοράς. Γι' αυτούς τους λόγους πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να, ελέγχονται, να ελέγχουν μάλλον και να καθορίζουν το επίπεδο συμμετοχής στις διάφορες δραστηριότητε. Σας ευχαριστώ. Σα uh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σημαντικό το θέμα και ο τομέας αυτό. Και η ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών είναι πολύ, πολύ σημαντικό θέμα. υπολογίζουμε 7 με 16% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Πολλά χρήματα ε, δηλαδή και πολλοί κόσμοι αποφεύγει για και, λόγους κέρδους κάποια πράγματα που αφορούν την φορολόγηση, την κοινωνική κάλυψη, οι κοινωνικές μηνυσφορές που όλοι θα πρέπει να καταβάλουμε. Τη στιγμή όπου ο δημο, το δημόσιο κορβαράς είναι τόσο πιεσμένος είναι πολύ καλή ιδέα. Βέβαια κάθε κράτος μέλος έχει τη δική του ευθύνη, αλλά η μοιρασιά των καλύτερων πρακτικών είναι πολύ καλή θετική και δεν είναι νέος τομέας όπως γνωρίζουμε για την έρευνα. Γίνεται εδώ και δεκαετίες από την Κομισιόν που προτείνει ε, ε, ιδέες. Μιλάμε εδώ για επιβολή του νόμου σε αυτή την Επιτροπή συχνά που είναι ακόμα ένας τομέας με δυσχέρειες και σίγουρα λοιπόν πρέπει να το διερευνήσουμε, να το στρίξουμε και οι κοινέ αρχές είναι κάτι που θα πρέπει να στηρίξουμε. Ευχαριστώ. Dennis, would like to come back on those points? Thank you. θέλεις να επανέλθεις? Ναι, μπορώ να είμαι σύντομος. Εγώ σέβομαι απόλυτα τις εθνικές ε, αρμοδιότητες. Δεν υπάρχει εδώ καμία παρεξήγηση. Νομίζω πως επίσης η Κομισιόν όταν ξεκίνησε αυτή την πρόταση πρόσεξε έτσι ώστε να σεβαστεί τις αρμοδιότητες αλλά Αν υπάρχουν ας πούμε μονομένα σημεία επαφή σε εθνικό επίπεδο όπως προτείνει η Κομισιόν και καποιοι κάτι μέλη που είναι όχι εμείς δεν θα το κάνουμε, τότε δεν λύνεται το ζήτημα της πρακτικής συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη, πράγμα που είναι απαραίτητο Πρέπει ίσως να γίνει σε διμερή βάση σε κάποιες ε, περιπτώσεις να δούμε ποιος είναι υπεύθυνο για να μην καταλήγουμε πάλι στο λάθος άνθρωπο. Δεν θα πρέπει να δίνουμε λαβή για τους ε, ε, όσους διαπράττουν αδικήματα γιατί αυτοί κερδίζουν από τη μη δεδηλωμένη εργασία. Ενιαίο λοιπόν σημείο επαφής αλλά και κάποια μορφή συμμετοχής Φαντάζομαι θα το συζητήσετε περαιτέρω οι σκιώδεις. Αλλά κάπου ενδιάμεσα ένα αριθμιστικό πλαίσιο δηλαδή και ένα σύστημα προαιρετικό είναι απαραίτητο για να, γίνει, για να γίνει, σημειωθεί εδώ πρόοδος. Βεβαίω, και ε, δεν θέλουμε να σπαταλήσουμε χρήματα χωρί λόγο, αλλά πρέπει να στηρίξουμε <coughs> την ε, πρωτοβουλία αυτή. Προσβλέπω στι ε, τροπολογίε σα και στην περαιτέρω συζήτηση του θέματο Και εγώ σα ευχαριστώ για τη συζήτηση. Το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι να ακούσουμε από την Κομισιόν τον κύριο Κέρτ Χάινεν για να απαντήσει στις ερωτήσεις για τις άδικες αθέμητες μάλλον πρακτικές ε, στην, ε, στην αλυσίδα των τροφίμων. Σας ευχαριστώ πολύ που επανήλθατε για να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Ο ε, συγητής μου έστειλε πολύ αργά χτες το βράδυ ένα μήνυμα όπου εξηγεί ότι έπρεπε να φύγει για την Πολωνία. At very late notice and Um, Τελευταία στιγμή και μου ζήτησε πολύ ευγενικά να σας, ε, σας πω ότι θα ακούσει τις απαντήσεις σας με μεγάλη προσοχή μέσω του βίντεο και ότι η βοηθό η βοηθός του είναι στην αίθουσα και θα συμπληρώσει και θα καταγράψει όλα τα σχόλια. Για το μέλλον λοιπόν, αν ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και θέλετε να σας να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματός σας σε, κάποια συνεδρίαση, ευχαρίστω να το κάνω για οποιονδήποτε από εσά. Η Κομισιόν λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να επανέλθω για τα πολλά ερωτήματα, τα χθεσινά. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με τη σειρά που μου ετέθησαν. Ξεκινώ λοιπόν με αυτά του εισηγητή, ο οποίος ανέφερε το φόβο Had, uh, how was to... και είπε πώς θα αντιμετωπίσουμε τον παράγοντα αυτό ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά τα εθελοντικά ε, σχήματα και προγράμματα, αν αυτό το παράγοντα μπορούν να τον αντιμετωπίσουν. Όπως ανέφερα στην εισαγωγή μου, ο παράγοντας ε, φόβος πραγματικά είναι ένα ζήτημα που βρίσκεται και στην καρδιά του όλου προβλήματος, της επιβολής. Διότι πράγματι έχουμε αυτές τις αθέμητες πρακτικές σε συμβατικές σχέσεις μακράς διάρκειας και το ένα συμβαλόμενο μέρος είναι εξαρτημένο ουσιαστικά από τη σχέση αυτή. Θέλει να συνεχιστεί αυτή η συμβατική σχέση. Και σε μια τέτοια κατάσταση είναι φυσιολογικό η αδύναμη πλευρά να έχει φόβο. Γι' αυτό και δεν προσφέρει. Είχαμε και την πράσινη βίβλο ηγητής. Και το θέμα αυτό το είχαμε θέσει, το λάβαμε και στις απαντήσεις μας στο πλαίσιο της εργασίας διαβούλευσης. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα αυτά τα εθελοντικά, ή αν όχι όλα με κάποια από τα εθελοντικά προγράμματα. Είναι ακριβώς αυτό ουσιαστικά. Η δυσκολία που υπάρχει. let's say, credible um, possibility. Δεν παρέχουν ουσιαστικά ε, τη δυνατότητα να υπάρχει και επιβολή αλλά και σεβασμός της εμπιστευτικότητας. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό στα συστήματα επιβολής να μπορεί κανείς να κάνει εμπιστευτικές καταγγελίες. και η αρχή ή οποιοδήποτε άλλος ασχολείται με τις καταγγελίες αυτές να μπορεί αυτεπαγγέλτος να προβαίνει σε έρευνα προστατεύοντας τον καταγγέλλοντα. Μάλιστα. Τώρα, η Κομισιόν καλεί τα κρατημέλη να το εξετάσουν αυτό στην ανακοίνωση. Επίσης, μάλιστα. Περνάω στην κυρία Σενάλοβα που ρώτησε το ότι οι αγρότες που δεν έχουν πει σε αυτήν την πρωτοβουλία τη αλυσίδα εφοδιασμού, πώ το αντιμετωπίζουμε και ότι είναι περιορισμένη η συμμετοχή των ΜΜΕ. εξέφρασε δηλαδή κάποιες επιφυλάξεις ό,τι αφορά ακριβώ αυτές τις θελοντικές πρωτοβουλίες. Πράγματι, είναι μια αδυναμία αυτής της πρωτοβουλίας ε, ελευθερίας εφοδιασμού, το ότι δεν έχουν ε, ενταχθεί αγρότες, το είπαμε και χθε και αυτό έχει να κάνει με το μηχανισμό επιβολής, αλλά ελπίζουμε και ξεκολουθούμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμη πιθανότητες να ενταχθούν και οι αγρότες σε αυτά τα θελοντικά συστήματα γιατί το βλέπουμε να γίνεται στις εθνικές πλατφόρμες. Συμμετοχή ΜΜΕ. Είναι μια ανησυχία για την πρωτοβουλία της αλυσίδας εφοδιασμού. Κάποιος πρέπει να είναι μέλος αυτής της πρωτοβουλίας για να μπορεί άμεσα να επωφεληθεί από αυτή την πρωτοβουλία. Βέβαια, πολύ σωστό και το επιχείρημα ότι εμέσως μπορούν και οι ΜΜΕ να ωφεληθούν από το γεγονός ότι αν οι μεγάλες εταιρείες εντάσσονται σε αυτήν την πρωτοβουλία και την εφαρμόζουν, αυτό ουσιαστικά θα πειράσει και τις πρακτικές τους, άρα εμέσως και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν στην αξιολόγηση που θα κάνουμε φέτος. Αλλά σας τα είπα και χθες αυτά. Υπήρξε ένα ερώτημα για τα περιθώρια των ε, λιανοπολιτών, πώς επηρεάζονται οι καταναλωτές, από αυτές τα θέματα της ε, πρακτικές κτλ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργεί ένα, έχει δημιουργήσει ένα εργαλείο για την παρακολούθηση των εξελίξεων των τιμών των τροφίμων, με στόχο να υπάρχει διαφάνεια. Βέβαια, δεν προσπαθεί να μετρήσει ακριβώς τα περιθώρια, αλλά να δει τι γίνεται με τις τιμές, πώς ε, μεταβιβάζονται στην αλυσίδα εφοδιασμού. Δεν έχουμε πλήρη δεδομένα. Αλλά σε κάποιο βαθμό υποθέτω ότι είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες για τα περιθώρια. Πώς επηρεάζουν οι θέσεις της τους καταναλωτές. Αυτό είναι δύσκολο να μετρηθεί. και δεν είναι και ο βασικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής. Βέβαια, θέλουμε και οι καταναλωτές να ωφεληθούν. Και αυτό θα γίνει αν η διαλυξίδα μου λειτουργεί σωστά. Τώρα έρχομαι στον κύριο Ροσφόρ που μίλησε για τις ε, διαφορετικές ε, δυνατότητε καταπολέμηση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών και μίλησε για το ενδεχόμενο ενός διαμεσολαβητή που θα είναι ο αρμόδιος. να εξασφαλίσει ότι είναι θεμητές πρακτικές που ακολουθούνται. Ίσως είναι μια πολύ καλή προσέγγιση. Χρησιμοποιείται σε ορισμένες δικαιοδοσίες, σε ορισμένες χώρες, όμως Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλές άλλες δυνατές προσεγγίσεις. Στη Γαλλία μάλιστα. Γίνεται εκεί ε, διαμεσολάβηση, υπάρχει το σύστημα της διαιτησίας και σε κάποιο βαθμό και ο αναθέτων adjudicator στην Αγγλία για τα προκριτικά έχει τις ίδιες αρμοδιότητες. Solution as flexibly as and as efficiently. Ο στόχος μας είναι να βρούμε την πιο αποτελεσματική μέθοδο. Μπορούμε δηλαδή να καταλήξουμε ενδεχομένω και σε συνδυασμό εθελοντικών και νομοθετικών πρωτοβουλειών. Όπου ο βασικό στόχος των θελοντικών πρωτοβουλειών είναι αν μπορούν τα προβλήματα να λυθούν με ευέλικτο τρόπο χωρίς αντιπαραθέσεις θα είναι και η προτιμητέα λύση. Νομίζω ότι ένα άλλο ερώτημα ήταν αν μπορούμε να έχουμε ένα κατάλογο αυτών των αθέμπτων εμπορικών πρακτικών. Κάποια κράτη-μέλη επέλεξαν την προσέγγιση αυτή. Και όχι τη θετική λίστα, τόσες καλές πρακτικές που επιλέγει η πρωτοβουλία. Το σημαντικό είναι να υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας. Γιατί αν έχουμε άκαμπτες λύσεις, αν έχουμε έναν άκαμπτο μαύρο κατάλογο, μια μαύρη λίστα, αυτή μπορεί να μην είναι και η καλύτερη δυνατή λύση. Γιατί και ακόμη και προσπαθεί να είναι πολύ ακριβής και συγκεκριμένος ο κατάλογος, επειδή έχουμε συνεχείς εξελίξεις και μεταβολές, δεν θα τα καλύπτει όλα. Μπορεί να προκύψουν και νέα φαινόμενα. Ο κ. Ντάντε τώρα ρώτησε για τις ε, εξελίξεις ιδιωτικό τομέα και για τις εκτινιατρικές πρακτικές. Παρακολουθούμε τι γίνεται και στον τομέα αυτό της εργασίας. certainly also. και βλέπουμε ότι υπάρχει και βελτίωση με τους information. Ε, καταναλωτές. Κάποιες φορές γίνεται, ε, έχουμε κάποιες καταχρήσεις, έχουμε κάποιες αθέμητες πρακτικές σε κάποιους τομείς. Βέβαια, ε, λένε οι καλές δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε με λάθος τρόπο τις επιστευτικές πληροφορίες. That um, DG Competition has recently um, made a, um, extensive study on... Έχει γίνει μια ιδιωτική, ε, έχει γίνει μάλλον συγγνώμη, μια μελέτη για την ε, καινοτομία, για την αλυσίδα τροφίμων. Ε, εκεί μελετήθηκε συγκεκριμένα το θέμα αυτό του δυτικού τομέα. Ελπίζω να έχω καλύψει τις ερωτήσεις που μου ετέθησαν χθε. Σα ευχαριστώ που μου δώσατε δυνατότητα να πάρω το λόγο σήμερα. Και βέβαια αν υπάρχουν ερωτήσεις ε, και σήμερα μπορώ ευχαριστώ να τις απαντήσω. Υπάρχουν δύο ευρωβουλευτές που έχουν ερωτήσεις. Η κυρία Σενάλοβα πρώτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις. Είχα και μία ερώτηση ακόμα για την εσωτερική αγορά και την περίπτωση που υπάρχουν πολυεθνικές οι οποίες μπορούν να εφαρμόσουν διαφορετικές πρακτικές σε διαφορετικές χώρες και θα ήθελα διευκρινήσεις παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το θυμήσατε, το ξέχασα. Λοιπόν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για εμάς, διότι και εμείς το εξετάζουμε από τη σκοπιά της εσωτερικής αγοράς, όπως είπα και χθες. Πολλές από αυτές τις αθέμητες πρακτικές γίνονται σε τοπικό επίπεδο. και μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε λοιπόν και σε τοπικό επίπεδο. Και φυσικά έχουμε επίγνωση ότι ενδέχεται να προκύψουν θέματα συντονισμού. Γιατί εντάξει, όταν τα κράτη-μέλη έχουν λύσεις για εθνικό επίπεδο, υπάρχει κατακαιρματισμός ανάμεσα στα διαφορετικά κράτη-μέλη και χρειάζεται συνδυασμός και συντονισμός. Αλλά πιο σημαντικό από το να έχουμε μία πλήρη εναρμόνιση είναι να μην υπάρχουν κενά στις εθνικές νομοθεσίες, και, γιατί αυτά δεν είναι παιχνίδια. Αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ, διότι φυσικά έχουμε δεχτεί και πάρα πολλή σχόλια για αυτή την άγρα δικαστηρίου, ανάλογα με, τις, με την νομοθεσία που μας συμφέρει. Και συνεχίζουμε λοιπόν να το εξετάζουμε. Υπάρχει επομένως αυτός ο κατακαιρματισμός. Από την άλλη, ίσως είναι υπερβολικό να εναρμονίσουμε αμέσως. Ίσως θα έπρεπε να προωθήσουμε μία ενημέρωση, μια καλύτερη ενημέρωση για να γνωρίζουμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές και από την άλλη να φροντίσουμε να διασφαλιστεί συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και να διασφαλιστεί επίσης ότι δεν αφήνουν κενά τα εθνικά συστήματα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Στάιλερ που ήρθατε εδώ. Είναι πολύ ευχάριστο που έχετε δυνατότητα να Μα δώσετε απαντήσει και λυπάμαι που δεν υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι εδώ. Σίγουρα θα με ενδιαφέρε να μάθω για, ε, για την εθελοντική προσέγγιση και την υποχρεωτική προσέγγιση. Να δούμε τι γίνεται εδώ. Διότι γίνεται όλο ένα και σημαντικότερο να εφαρμόσουμε σωστά τα μέτρα και εσείς μας είπατε για την επιβολή και την εφαρμογή και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, το συζητάμε πολύ εδώ στην Επιτροπή. Από ό,τι καταλαβαίνω είστε επίσης αρμόδια για την ομάδα υψηλού επιπέλθου για το λιανικό εμπόριο. Και σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα στο λιανικό εμπόριο διότι αποτελεί το κύριο παράδειγμα όσων συζητούμε εδώ. Θα ήθελα λοιπόν να με ενημερώσετε για αυτό το θέμα, να μου πείτε αν το λιανικό εμπόριο περιλαμβάνεται στις συζητήσεις σας και το τι γίνεται με αυτό. Και επίσης τι επικοινωνία υπάρχει με τους οργανισμούς ε, Fair Trade για το δίκαιο εμπόριο. Διότι είχαμε και κάποιους προσώπους αυτή την εβδομάδα εδώ. Μάλιστα. Δημιουργήσαμε αυτήν την ομάδα υψηλού επίπεδου για το λιανικό εμπόριο. Ήταν μέρος του σχέδιου δράσης για τη λιανική που ετέθησε ισχύ το 2013. Και επίσης ήταν μέρος και του σχεδίου για τις ε, δικές εμπορικές πρακτικές. Η ομάδα υψηλού επίπεδου για τη λιανική δεν αστίασε τόσο πολύ στις δικές εμπορικές πρακτικές, γιατί Είχαμε θέμα χρόνου. Ήταν, ήρθε η ανακοίνωση τον Ιούλιο. Έπρεπε μετά να αξιολογήσουμε αυτά τα εθελοντικά προγράμματα και το πώς λειτουργούν στα κράτη-μέλη και δεν ήταν λοιπόν ένα θέμα που εξέτασε το... η ομάδα υψηλού επίπεδου. Η κύρια πρόκληση που εντόπισε η ομάδα υψηλού επίπεδου για το ελληνικό εμπόριο ήταν η ψηφιακή μεταρρύθμιση του τομέα, η ψηφιακή μεταμόρφωση, ψηφιοποίηση αν θέλετε και η σύνδεση αυτής της ε, αλλαγής με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως σας είπα λοιπόν, δεν ήταν ένα από τα κύρια θέματα που απασχόλησαν την ομάδα υψηλού επίπεδου και ένας από τους λόγους, όπως σας είπα, είναι και ο χρόνος, γιατί πραγματικά βρισκόμαστε σε μια φάση που περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα του εθελοντικού προγράμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. και πώς η εθνική νομοθεσία αντιδρά και πώς εφαρμόζεται και τι προβλέπει. Γι' αυτό πιστεύω πως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να το κοιτάξουμε αυτό. Πρώτα πρέπει να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν φέτος και μετά να επαναξιολογήσουμε τις ε, θεμητές εμπορικές πρακτικές. Σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα θα έχουν και άλλες ερωτήσεις τα μέλη της Επιτροπής κατά τη διάρκεια σύνταξης της έκθεσης. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και τις συμβουλές σας για το θέμα αυτό. Και θα είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πρέπει να πω επίσημα ότι η επόμενη συνεδρίαση θα αρχίσει στις 9 η ώρα το πρωί την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.